Συνάδελφοι, καλημέρα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που δεν έχω συναντήσει ήδη, αλλά ε, ευχές για ένα καλό νέο έτος, 2020, και για μια δραστήρια χρονιά στην Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αιτήματα για αλλαγέ, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί. Ευχαριστώ. Και τώρα μια ανακοίνωση σε σχέση με το Brexit. η σύνθεση του Κοινοβουλίου θα αλλάξει λόγω τη αποχώρηση του ΕΒ. Βασιλείου. Το γνωρίζετε. Έχουν ληφθεί οι απαραίτητε αποφάσει στην προηγούμενη Ολομέλεια. Για τη δική μα την υποεπιτροπή δεν θα υπάρχουν αλλαγέ σε σχέση με τον αριθμό των τακτικών μελών. Θα είμαστε 30. Τέσσερι ε, Βρετανοί συνάδελφοι μα αφήνουν. Δύο τακτικά μέλη, ο κ. Φαν Όρνταν και ο κ. Μπράι. Και δύο αναπληρωτέ. Hollywood και Θα ήθελα λοιπόν επειδή θα φύγουν, να χαιρετήσω τη συμβολή τους στις εργασίες αυτού του Κοινοβουλίου και στις ονοματοτήσεις αυτού του Κοινοβουλίου. Θέλω να τους πω ότι για μας είναι δυστυχώς ε, ατυχές το ότι φεύγουν. Χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι πια ίδια. Και τους εύχομαι ε, κάθε τύχη στην επαγγελματική και προσωπική τους ε, πορεία για το μέλλον. Να σας θυμίσω επίσης ότι η κυρία Ισουμίνα Κανίτσου, η οποία είναι ε, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα θέματα του αφοπλισμού, μας έκανε την τιμή να δεχτεί την πρόσκλησή μας και να συμμετάσχει σε μία συνεδρίαση 27 ε, Ιανουαρίου της Υποεπιτροπής αυτής, 27 Ιανουαρίου, ε, ευκαιρία να έχουμε διάλογο με την κυρία Νακαμίτσου για την συνθήκη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και την διαδικασία παρακολούθησης της στήρισής της. Και θα ασχοληθούμε γενικότερα με το θέμα αυτό, με τη συνθήκη. Περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, 12 Νοεμβρίου, 21 Νοεμβρίου, 2 και 3 Δεκεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Και τώρα περνάμε στο σημείο 4. Ανταλλαγή απόψεων για τι στρατιωτικέ προκλήσει στην περιοχή του Σαχέλ, νοτιό τη Σαχάρα. Το έχουμε προβλέψει σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω του ομιλητέ μα. Όλο ιδιαίτερο τον κύριο Έσα Πουλκίνεν, Γενικό Διευθυντή του Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κυρία Μπριγκίτα Μάρκουσεν, Γενική Διευθύντρια, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για την Αφρική στο ΣΕΑΕ και τον αντινάβαρχο Ξαβιέ Πετή, που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ε, διοικητική μερίμνα στι επιχειρήσει, στο κέντρο σχεδιασμού επιχειρήσεων και την διεξαγωγή των επιχειρήσεων στο επιτελείο του Γαλλικού στρατού, καθώ και τον κύριο Ρέκαν, ο οποίο είναι ε, αποσπασμένο ε, του Εστονικού αμυντικού μηχανισμού στην Γαλλία. Ε, κάποια λόγια εισαγωγικά. Στις 11 Ιανουαρίου 2013 η Γαλλία ξεκίνησε την επιχείρηση Σερβάλ με 1.800 στρατιώτες για να σταματήσει την πρόοδο των τζιχαντιστών που ήλεγχαν τον βορρά του Μάλι και να υποστηρίξει τα στατεύματα αυτής της χώρας από την απειλή κατά της πρωτεύουσα Μπαμάκο. 1η Αυγούστου 2014 η επιχείρηση αυτή καταστάθηκε από την επιχείρηση Μπαρκάν, η οποία ε, διευρύνθηκε στο σύνολο της ζώνης νοτίως της Σαχάρας στο Σαχέλ. Η... Ο ΙΕ δημιούργησε το ΣΥΝΟΣΜΑ ε, 16.000 στρατιώτες για να υποστηρίξει την ε, κρατική αρχή στα βόρεια του Μάλι. Από το 2013 η απειλή ε, κατά ε, από την διχαντιστική τρομοκρατία έχει προχωρήσει. Ξέρουμε ότι έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπλώνονται σε πέντε χώρες του Σαχέλ. Και σήμερα στο Μάλι ε, την επιχείρηση Μπαρκάν ε, χειρίζεται η Γαλλία με συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Εστονίας, της Δανίας και η επιχείρηση του ΙΕ όπου υπάρχει συμμετοχή ε, παρακολουθείται από τις χώρες του G5. Έχουν διοργανωθεί λοιπόν δύο επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι με 22, χρόνια, με 22 χώρες να εκπροσωπούνται και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσα στρατεύματα ε, με τόσες χώρες παρούσες θα έπρεπε να επιτρέψουν στις καθηγές αρχές, στις νόμιμες αρχές να ξαναπάρουν τον έλεγχο της χώρας. Όμως υπάρχουν τραγικές απώλειες που ε, ε, δικαιολογούν τη σημερινή εξέταση του θέματος ε, καταλεπτός κιόλας. Μάλιστα, στο ΠΟ στη Γαλλία στις 13 Νοεμβρίου διοργανώθηκε σύνοδος που επιβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή και διεθνής παρουσία στο Σαχέλ, νοτίος της Σαχάρας, είναι νόμιμη βάση του αιτήματο των χωρών της περιοχής και από τη μια, ε, η σύνοδο επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης της Διεθνού και ευρωπαϊκής παρουσίας στα πλευρά στο πλευρό των συμμάχων μας του G5. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στην κυρία Μάρκουσον ε, για να μας κάνει μια ε, ανακεφαλαίωση του πώς έχουν τα πράγματα στο Σαχέλ και σε σχέση με την κατάσταση της ασφάλειας. Τα πράγματα μα ανησυχούν. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώ προχωρούν οι κινήσει τη διεθνού κοινότητα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα την εισήγηση αυτή να την κάνω επικεντρωνόμενη σε τέσσερα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, η συνολική αποτίμηση ασφάλειας ε, της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της μετά δύο σομαριτικές συναντήσεις, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα αυτή την εβδομάδα που συζήτησα για το Σαχέλ και όπως είπε και η Πρόεδρος, η συνάντηση στο ΠΟ. Ε, και μετά έχω κάποια συμπεράσματα για το πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα εξετάσουμε το θέμα αυτό. Τώρα, τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν τα θέματα του Σαχέλ. Ήδη από πέρσι είχαμε μια εντατική πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο και πέρσι το Μάιο είχαμε μια σωρία συνεδριάσεων με υπουργού εξωτερικών, μετά με υπουργού άμυνα που έχουν σχέση με την Επιτροπή σα και μετά μεταξύ των Υπουργών Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Οι εντατικές αυτές διαπραγματεύσεις πέρσι γίνονται στα πλαίσια μιας θλιβερής παναχώρηση. Είδαμε χθε μόλις το βράδυ να έχουμε νέες επιθέσεις ε, κατάμαχων, 30 τουλάχιστον νεκροί στην Πουρκίνα Φάσο. Εάν δούμε τους αριθμούς που έχουμε μπροστά μας, οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν οδηγήσει στο θάνατο 1.500 Αφρικανών στρατιωτών και αν αρχίσουμε να μετράμε και άμεχου πολίτε, φτάνουμε του 4.000. Είναι ανησυχητική η αριθμή, είναι σοβαρό το θέμα ασφάλεια, αλλά βλέπετε και τι συνέπειε υπάρχουν από τι πολιτικέ κινήσει και αποφάσει εδώ. Ε, άρα ήταν σημαντικό να συναντηθούμε στο ΠΟ, θα σας ενημερώσω για τις σχετικές εξολήξεις και στο Βόρειο Τσάντ. Θα συναντηθούν οι πέντε χώρες του Σαχέλ τέλη Φεβρουαρίου, είναι και αυτό σημαντικό και μετά να πω ότι αυτή τη στιγμή οργανώνουμε συνάντηση ανώτου του επίπεδου ταυτόχρονα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 26 Μαρτίου εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα συμπεράσματα από την τώρα προσπάθειά μας και από τη σύνοδο του ΠΟ δείχνουν τα εξής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι εφόσον θέλουμε να εντατικοποιήσουμε την παρουσία μας στο Σαχέλ πρέπει να έχουμε μια ενοποιημένη προσέγγιση πολύ συχνά μιλάμε για έναν άξονα, δεν είναι όμως έτσι. Πολιτικός, διπλωματικός, ε, ασφάλειας και άμυνας, αυτοί οι άξονες πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. Και ο ανθρωπιστικός και ο αναπτυξιακό. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πέμπτο άξονα, Υπάρχουν χώρε που θα ήθελαν και οικονομική δραστηριότητα, αλλά αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι σημαντικό λοιπόν για μα να δείξουμε ότι υπάρχει ενωπημένη προσέγγιση εδώ, μια ημιογενή προσέγγιση, διότι τα πράγματα στην πράξη δεν θα επιληθούν μόνο με στρατιωτικά και αμυντικά μέσα, αλλά υπάρχει και ανθρωπιστική κρίση και ε, χρειάζονται προσπάθειε αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό που ξέρουμε όμω τώρα, εξετάζοντα την κατάσταση, είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το Σαχέλ και αυτό θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί σήμερα. Τρία είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να ξαναδούμε διαφορετικά τα πράγματα σε συνδυασμό και με την ε, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών αυτή την εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κινητοποιήσουμε τον πολιτικό πυλώνα, να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες να κοιτάξουμε να πετύσουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις. Βεβαίως, οι χώρες αυτές είναι πολύ φτωχές, έχουν λίγες δυνατότητες. Όμως, εάν δούμε την ηγεσία των πέντε χωρών, μπορεί κανείς να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα, να καταλάβει το ρόλο της πολιτικής ηγεσία. Είναι σημαντικό. Επίσης, θέλουμε η αναπτυξιακή μας συνεργασία να είναι πιο στοχευμένη, να παρακολουθούμε ακριβώ πού πηγαίνουν τα κονδύλια χρειάζονται αμοιβαίε δεσμεύσει για το πώ εργαζόμαστε, για τα αποτελέσματα που απαιτούμε και τι μεταρρυθμίσει που θέλουμε από τι συγκεκριμένε χώρε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, είναι ότι πρέπει να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας ξανά στο γεγονός ότι τα κατεπήγοντα και τα πρόβλεπτα είναι η κανονική κατάσταση σε αυτή την περιοχή πλέον και πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη νέα κατάσταση. Ξαναμελετούμε τους τέσσερις άξονες που σας είπα προηγουμένως, πολιτική, ασφάλεια, ανάπτυξη, ανθρωπιστικά, αλλά η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι εντελώ έκτακτη. Γι' αυτό η σύνοδος ε, των G5, των χωρών G5 τέλη Φεβρουαρίου, θα μας δώσει ε, ένα σφιγμό. Ε, τη κατάσταση ε, πέρσι ανέπτυξαν ένα ενοποιημένο πλαίσιο. Ε, συμφωνήσαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε ευπαθεί περιοχέ σε κάθε μια από τι πέντε χώρε. Χρειάζεται τώρα μια πιο ομοιογενή προσέγγιση. Λίγα λόγια για τη σύνοδο του ΠΟ τη περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα. Ήδη το είπα, αυτή τη συλλογιστική ακολουθήσαμε βάσει των τεσσάρων αξώνων. Αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, στρατιωτικέ επιχειρήσει, πρώτο άξονα μετά αμυντική ε, οργάνωση, μετά ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού, των κρατικών μηχανισμών και μετά ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι σημαντικό οι διάφορες πρωτοβουλίες που υπάρχουν και είναι πολλές να οργανωθούν οριζόντια, εγκάρσια μάλλον, ε, και αυτό πρέπει να συντονίσουμε. Το τελευταίο, και εδώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω, γιατί θέλω να έχουμε χρόνο και για συζήτηση, από την σκοπιά των Υπουργών Εκτορικών και από την ΕΕ τα κράτη-μέλη θέλουν περισσότερη και εντονότερη ε, δέσμευση, ανάληψη δράσης για το Σαχέλ. Πρέπει επίσης να δούμε τα πορίσματα της Συνόδου του ΠΟ από τη Γαλλία και τους τέσσερις πυλώνες που σας περιέγραψα, να τους αξιοποιήσουμε και μετά Υπάρχουν αρκετά κρατημέλη που είναι τη άποψη ότι χρειάζεται ενισχυμένη και ε, εκτεταμένη πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε τις θετικέ αναθεωρήσεις σε αυτό το πλαίσιο, αυτές που τώρα προγραμματίζουμε, και μετά η σφαιρική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σοβαρότατη κρίση που έχει προκαλέσει πολλούς νεκρούς ε, και αμάχους και στατιώτες. Υπό αυτή την έννοια προετοιμαζόμαστε και για τη σύνοδο της 26ης Μαρτίου. Κάνουμε τώρα ό,τι μπορούμε και αναλύουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της ασφάλειας, τι χρειάζεται για τη σταθεροποίηση και πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα χάσματα στην Σύνοδο του Μαρτίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Μιλήσατε λοιπόν για τις επόμενες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αντιστράτηγο Πιουτίνεν, Πούλκινεν, ο οποίος θα μας μιλήσει για το μαλή 14.000 στρατιώτες του Μαλί ε, ε, έτυχαν εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένας τεράστιος αριθμός. Βέβαια, ο ποσοτικός στόχος δεν αρκεί. Η εντολή είναι το θέμα και οι απαραίτητες προσαρμογές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να βοηθούμε τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλή να είναι έτοιμες, να παρέμβουν, να είναι λειτουργικές και να μπορούμε να τους πλαισιώνουμε όσο δυνατόν πιο κοντά επιτόπου. Συνδέοντας την επιχείρηση Μπαρκάνα με μια ιδιαίτερη προσπάθεια στο κέντρο του Μαλή τίθεται όλα αυτά τα ζητήματα επιτάπητο σήμερα και αντιστράτηγε κοινέν θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μάθουμε ποια είναι η κατάσταση αλλά και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Σας ευχαριστώ και σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση που μου απευθύνεται να εκφραστώ ενώπιον της Επιτροπής σας. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνομιλώ με τους αιρετούς εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Είχα έρθει και πριν από δύο εβδομάδες για να τοποθετηθώ για κάποια άλλα ζητήματα, γιατί είναι δύο οι βασικές μου ιδιότητες. Είμαι ο στρατάρχης επικεφαλής του επιτελείου και ε, συνομιλώ με, ε, για θέματα στρατηγικά ε, για θέματα πολιτικής προστασίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι και επικεφαλής της εκπαίδευσης της στρατιωτικής που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες ενοπλές δυνάμεις άλλων τρίτων χωρών στην Αφρική. Θα ήθελα λοιπόν να, να μιλήσω και με τις δύο αυτές ιδιότητες. Συμφωνώ απολύτως με την προλαλήσασα ε, για την κατάσταση. Έτσι έχει η κατάσταση και έτσι είναι και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ενοποιημένη, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε, ε, το στρατιωτικό σκέλος ε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αλλά αυτή η συμβολή δεν λαμβάνει χώρα εν κενό. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, αυτό είναι προφανές και δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε αυτή την ενοποιημένη, την ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, ε, με τα Ηνωμένα Έθνη, με τη Γαλλία, με τις μεγάλες χώρες και με κάποιες χώρες τις οποίες αποκαλούμε οι ντόπιοι φίλοι μας. Okay, Υπήρξε μια τεχνική διακοπή, μια έξωθεν παρέμβαση. Από στρατιωτική σκοπιά, αν δείτε τη Δυτική Αφρική, είναι μια ενιαία ε, γεωγραφική περιοχή στην οποία παρεμβαίνουμε από τον κόλπο της Γουινέας μέχρι το Μαλί, τη Δυτική Λιβύη και τη Μεσόγειο. Είναι μια ενιαία στρατιωτική ε, προοπτική. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή αυτή τη τεράστια περιοχή ως ε, ένα σύνολο γεωγραφικό. Έχουμε τον τζιχαντισμό, ο οποίος επικρατεί, ο οποίος συνεχώς αυξάνει τις δυνάμεις του. Όχι μόνο στο Μαλί, αλλά και στην Μπουρκίνα Φάσο και στον Νίγηρα και σε άλλες χώρες. Αυτή είναι μια διάσταση η οποία πρέπει κάτι να γνωρίζει και είναι εξαιρετικά σημαντική. Ένα άλλο στοιχείο αστάθειας προκύπτει από το γεγονός ότι σημειώνονται εθνοτικής φύσης συγκρούσεις οι οποίες εξελίσσονται και αυξάνονται. Στο κέντρο του Μαλή συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που σχετίζονται με το εξωτερικό, με τις άλλες χώρες, αλλά έχουν και την εσωτερική τους δυναμική στο εσωτερικό της χώρας και εξελίσσονται και ανεξάρτητα. Πριν από λίγε μέρε ως προς τη στρατιωτική αποστολή εκπαίδευση. πρέπει να σας πω ότι κλείσαμε τα 7 χρόνια κατά τα οποία εκπαιδεύουμε στρατιωτικά τις ενόπλε δυνάμει. Και αν ε, δεν απατώμε, ο ε, ο, ο Γάλλος Γεθά αυτή τη στιγμή ε, ήταν ο πρώτος επικεφαλής της ε, εκπαιδευτικής στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή πριν από 7 χρόνια. Είναι διαφορετικές ε, οι εντολές της στρατιωτικής εκπαίδευσης και διαφορετικές εντολές της μηνούσμα, της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς δεν φέρουμε όπλα, έχουμε ισχυρή προστασία βέβαια όμως ο ρόλος μας είναι καθαρά ή περισσότερο, αν θέλετε, εκπαιδευτικός, συμβουλευτικός και ένας ρόλος δηλαδή ε, του να είμαστε οι πνευματικοί πατέρες και να καθοδηγούμε τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας. Συνεχίζουμε τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να έχουμε ένοπλες δυνάμεις στο Μαλί που να μπορούν να επιβιώσουν, που να μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου, να χαρακτηρίζονται από αηφορία δηλαδή συμβουλεύουμε και για ε, τη χρηματοδότηση και για τον εφοδιασμό και την ε, επιμελητεία και για τη στρατολόγηση, την τοπική πολιτική στρατολόγηση. Δεν κάνουμε μόνο εκπαίδευση σε ανθρώπους, ε, στρατιωτική εκπαίδευση σε ανθρώπους, αλλά συμβουλεύουμε για το πώς θα μακροημερεύσει και θα επιβιώσει και θα ευημερήσει ο Εθνικός Στρατός, οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας αυτής. Τις ένοπλες δυνάμει της απασχολεί κυρίως η αυξανόμενη αστάθεια στο κέντρο του Μαλή και υπάρχουν επιχειρήσεις στρατιωτικέ, εξαιρετικά βαριέ, επαχθεί, επίπονες και άρα είναι δύσκολο εμείς ε, να κάνουμε την εκπαίδευση για τον στρατό σε καιρό ειρήνη, σε καιρό μη εμπόλεμων ε, συγκρούσεων και για το πώς θα οργανωθεί καλύτερα. Στον Παμάκο έχουμε κάνει δραστηριότητες εκπαιδευτικές και θα ξεκινήσουμε και αντίστοιχες δράσεις στο Τιμπουκτού, αρκετά μακριά, στα βορειοανατολικά της χώρας, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικές μας δράσεις να απλωθούν στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας. Σε δεδομένες βέβαια συνθήκες και καταστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Στη στρατιωτική κοινότητα η συζήτηση στρέφεται κυρίως γύρω από το πώς θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μας αποστολής. Σε αυτό το πλαίσιο κατά το οποίο η εντολή μας είναι μη εκτελεστική. Και αυτή είναι η ουσία των στρατιωτικών επιπτώσεων της ε, στρατηγικής μας θεώρησης και αντιμετώπισης ε, και αναθεώρησης της κατάστασης σε σχέση με το κέντρο του Μάλι. Εμείς κάνουμε τη στρατηγική αναθεώρηση και θα την παρουσιάσουμε στην αρμόδια επιτροπή. Τονίζουμε την ανάγκη να είμαστε παρόντες μόνιμα, σε με πιο μόνιμο χαρακτήρα. Και υπάρχει διάταξη να ε, στηρίξουμε τις τοπικές δυνάμεις των ε, χωρών ε, G5. Μιλούμε για μια έκταση 5 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, τη μισή Ευρώπη δηλαδή. Και περιλαμβάνεται εκεί και το θέμα της Μπουρκίνα Φάσο. Όλα αυτά είναι στην εντολή μας. Συμφωνώ με τις φιλοδοξίες σε υψηλού επίπεδου. Πρέπει να έχουμε μια πιο μόνιμη παρουσία, αλλά εξαρτώμαστε και από τα κράτη-μέλη και από τη βούλησή τους να εμπλακούν, να συμμετάσχουν και να μας δώσουν τους απαραίτητους ανθρωπίνους πόρους να μας δώσουν ε, τη στήριξη σε θέματα εφοδιασμού, επιμελητίας, αερομεταφορών, η ε, ατροφαρμακευτικης περίθαλψης. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή. και πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Δεν μπορέσαμε να στρατολογήσουμε αρκετούς ανθρωπίνους πόρους, γαλλόφωνους, αξιωματικούς κυρίους. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο ενεργητικού, το βασικό προσόν για να μπορέσουμε να συμβουλεύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλή. Και υστερούμε και στις ιατροφαρμακευτικές μας δυνατότητες και στις αερομεταφορές. Φαίνεται ότι επιλέγουμε συνεχώς λύσεις υπεργολάβων και ανάθεση σε τρίτον, γιατί τα κράτη-μέλη δεν δίνανται να μας δώσουν, να μας καλύψουν αυτές τις ανάγκες, το οποίο δεν είναι και βέλτιστη λύση. Θα ήθελα όμως να ολοκληρώσω εδώ την ε, παρέμβασή μου, λέγοντας ότι η Αφρική είναι πολύ σημαντική για εμάς. η Δυτική Αφρική, η ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ. Κάνουμε μια επένδυση σε βάθος χρόνου, η οποία δεν είναι μόνο επένδυση για την Αφρική, αλλά είναι επένδυση και για τα δικά μας παιδιά εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε υπομονή, δεν μπορούμε να τα πετύχουμε σε μια-δυο μέρες. Μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες. Είναι μια επένδυση όμως που θεωρούμε ότι θα αποδώσει ε, σε βάθος χρόνου και για την Αφρική και για την Ευρώπη. Επίσης, από την πολιτική σκοπιά τίθεται θέμα στρατηγικής ε, και στρατιωτικής αυτονομίας της Ευρώπης. Είναι ευθύνη της Ευρώπης να φροντίσει την Αφρική, κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει, εμείς πρέπει να το κάνουμε και θα είναι ε, και μια δοκιμασία πολύ σημαντική για τα επόμενα χρόνια. Εάν καταφέρουμε να φροντίσουμε την Αφρική μαζί με τους Αφρικανούς φίλους μας, θα αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να φροντίσουμε για τη δική μας ασφάλεια και να εγγυόμαστε για τη δική μας ασφάλεια σε βάθος χρόνου. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την ενηλικίωση της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον Αντινάβαρχο Πετή. Νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής ενδιαφέρονται να ακούσουν τις ε, απόψεις σας για την επιχείρηση Μπαρκάνε και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και τις προοπτικές για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την επιχείρηση στο Σαχέλ. Όπως ξέρετε, η επιχείρηση Μπαρκάνε προέρχεται από αίτημα των χωρών του Σαέλ υπάρχει από το 2013 που από το 2013 και μετά δεν μπορούσαν να ελέγξουν τόσο την περιοχή και την εξέλιξη, οπότε χρειάστηκε, χρειάστηκαν βοήθεια για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών ομάδων επιτόπου. Ο αντίπαλος είναι ένα μοσαϊκό διαφορετικών οργανώσεων με διαφορετικούς στόχους και αιτίες προέρχονται από παλαιές αντιπαλότητες, ε, εθνοτικές διαφορές και οικονομικές δυσκολίες. Παροτρύνονται και από θρησκευτικέ διαστάσεις και από εξωτερικούς υποστηρικτές. Συνδέονται με το al ή το al με βάση συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον κόσμο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αν μπορέσουν θα επεκταθούν σε, όλη την περιοχή, ιδίως στις χώρες του νότου του κόλπου της Γουινέας, ε, Κόγκο, Ακτή, Φαντοστού, Μπενέν κλπ. Δημιουργώντας ένα χαλιφάτο με πιθανή δυνατότητα ευρύτερη δράσης τους αργότερα στην Ευρώπη, όπως είδαμε στη Μέση Ανατολή. Ήδη οι τρομοκράτες αποσταθεροποιηθούν τα κράτη και τους πληθυσμούς της περιοχής, τα σχολεία κλείνουν, οι δημόσιες υπηρεσίες ε, ε, εξαφανίζονται, δολοφονούνται πολίτες. Ε. Στρατιωτικά είναι δύσκολο να χτυπήσουμε τον εχθρό αυτό γιατί λειτουργεί με ασύμετρο τρόπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να σέβεται το δίκαιο των ενόπλων σειράξεων, κρύβεται μέσα στον πληθυσμό, ιδίως μέσα σε ένοπλες ομάδες που είναι εξουσιοδοτημένες να φέρουν όπλα έχουν την υποστήριξη του ντόπιου, κάποιου μέρους του ντόπιου πληθυσμού γνωρίζουν την περιοχή, γνωρίζουν πού μπορεί να κρυφθούν εύκολα, ιδίως στις περιοχές του κέντρου, που δεν είναι όπως φαντάζεται κανείς μια τεράστια έρημος, είναι δασωμένη περιοχή, Άρα ο εχθρό μπορεί κάλλιστα να κρυφτεί σε κάποιες περιοχές εύκολα. Είναι δύσκολο να τους βγάλουμε από τις, τα κρυσφύγετά τους. Μπορούν να ζήσουν στην έρημο, να ενταχθούν στον τοπικό πληθυσμό χωρίς, μέτρα, χωρίς με πολλά μέσα, χωρίς υποστήριξη. Χρησιμοποιούν το ίντερνετ, το τηλέφωνο drones, ε, μικρά προϊόντα με αποδεδειγμένη ωστόσο ε, ικανότητα. Η επιχείρηση αυτή έχει στόχο να επιτρέψει στις χώρες του Σαχέλ να ε, αντιμετωπίσουν με αποφασιστικό τρόπο την κατάσταση. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να χτυπήσουμε άμεσα τους τρομοκράτες, να αντιμετωπίσουμε τα δίκτυα, την ηγεσία τους και να υποστηρίξουμε τους εταίρους μας ώστε αύριο να γρήγορα δηλαδή να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτή την τρομοκρατική ε, απειλή με ένα πιο στεναρό τρόπο που θα μπορεί να επιτρέψει στα κράτη να αντιμετωπίσουν ευθέως την τρομοκρατία. Η ζώνη δράσης της επιχείρησης Μπαρχάν εκτείνεται σε μια επιφάνεια 10 φορές μεγαλύτερη από τη Γαλλία, σαν την Ευρώπη σχεδόν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεγάλος μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Εμείς έχουμε 4.500 ε, στρατιώτες αυτή τη στιγμή. Το κέντρο, βρίσκεται, το κέντρο δράσης βρίσκεται στην Τζαμένα με επικεφαλής μια δομή που στηρίζεται στην Μετρόπολη και εξασφαλίζει τον έλεγχο της αεροπορίας ε, που έχει κέντρο στο, στη, στη Λιόν. Η υποστήριξη, η αεροπορική υποστήριξη επιτρέπει αυτόνομες βράσεις της ε, ομάδα του, του, του στρατιωτικού αυτού οχήματος βορρά και νότου. Στην Τζαμένα υπάρχει και ε, η διοίκηση και μια στρατιωτική και μια αεροπορική παρουσία με, με υποστήριξη και μεταφορική και υποδομών. Στο δυτικό κομμάτι, στο Μαλί κυρίως, έχουμε δύο ομάδες στρατιωτικού προσωπικού με υλικό όπως οχήμα, ε, οχήματα, μία, ένα, μία ομάδα ε, ελικοπτέρων, μεταφορικών και επιθέσεων. Η γαλλική παρουσία συμπληρώνεται από την παρουσία μιας ομάδα 50 περίπου Εσθονών, Βρετανών, ελικόπτερα 1647, Ισπανικών δυνάμεων ε, με τακτική και, ε, στρατιωτική μεταφορά, υποστήριξη της Γερμανίας που κάθε, ε, κάθε εβδομάδα παρέχει κάποιες πτήσεις στην περιοχή, δανική υποστήριξη που παρέχουν δύο ελικόπτερα και η αμερικανική υποστήριξη μέσω στρατηγικών μεταφορών και παροχής πληροφοριών. Αυτό είναι η, άμεση υποστήριξη στην επιχείρηση Μπαρχάν. Θα μιλήσω αργότερα για τις διάφορες άλλες ε, Πρόκειται λοιπόν για σημαντική δράση για να εξουδετερωθούν οι τρομοκράτες με διάρκεια, όχι μόνο για ένα μικρό διάστημα. Η δράση γίνεται στο κέντρο της περιοχής του Μαλή και κοντά στο Νίγηρα, κοντά στην Κόρμα, στην Κούρμα, δηλαδή σε περιοχές ε, που είναι το τριεθνές μεταξύ Μαλή, Μπουρκίνα, Φάσο και Νίγηρα την περιοχή δηλαδή της ε, βασικής παρέμβασης της τρομοκρατίας. Όπως αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΠΟ, ο πρόεδρος ε, Μακρόν αποφάσισε να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία ενώ όπως αναφέρθηκε οι τρομοκράτες συνεχίζουν να επιτίθενται και να διευρύνουν τις δράσεις τους προς τα νότια, προς τον Μπουρκίνα Φάσο. Αποφασίσαμε λοιπόν ενίσχυση προσφέρθηκαν 220 ε, στρατιωτικοί στην ομάδα και δώσαμε μία υποστήριξη με την Task Force Takuba, μια επιχείρηση δυνάμεων που επιτρέπει να στηρίξουμε το Μαλί στην περιοχή του Λίτακο, κοντά δηλαδή στην περιοχή του Τριεθνούς που προανέφερα. Συνεχίζοντας την περιγραφή των μεθόδων δράσης μας, βρισκόμαστε σε συμβίωση με τις δυνάμεις της Μίνουσμα, το, της ομάδας των πέντε για το Σαχέλ και στόχος μας είναι ο έλεγχος της περιοχής και η συνέχιση της επιχείρησης Μπαρχάν, ιδίως στο πλαίσιο του αφοπλισμού που θέλουμε να ε, εξασφαλίσουμε κατά βάση μέσω της μήνουσμα. Η εμπλοκή του ΟΗΕ είναι σημαντική γιατί η περιοχή είναι τεράστια. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα έδαφος τόσο εκτεταμένο με μια μικρή ομάδα. Μαζί με τον Μπαλκάν λοιπόν υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή και αυτό είναι και αυτός ήταν και ο στόχος της ε, συνόδου του ΠΟ να ενισχύσει αυτή τη συμμαχία των ένοπλων δυνάμεων που έχουν εμπλακεί εκεί. Ε, η δραστηριότητα γίνεται με την ομάδα των πέντε του Σαχέλ, είναι η ελπίδα μας για το μέλλον, ενισχύεται ε, από τις πέντε χώρες του Σαχέλ που ε, από το 2014 και μετά συνασπίστηκαν για να αντιμετωπίσουν από κοινού την τρομοκρατία, δημιούργησε μια κοινή δύναμη που ενισχύεται τον τελευταίο καιρό και έχει προσπαθεί να φτάσει σε ένα στόχο 5.000 ατόμων, ενισχύοντας και τη μορφή των δράσεων που υλοποιεί. Έχουμε έξι επιχειρήσεις ε, στην περίοδο 2017-2018 ενώ το 18-19 η ποιότητα έχει αυξηθεί σημαντικά των, των αποτελεσμάτων και οι προσπάθειες της ομάδας αυτής έχουν σαν τελικό στόχο να μπορούν να επιλύσουν μόνες τους το πρόβλημα. Υπάρχει μια βούληση υποστήριξης από μας και γι' αυτό η Μπαρχάν ακολουθεί από δίπλα, δηλαδή στην ουσία λειτουργεί σαν ένας μαγνήτης των δραστηριοτήτων της ομάδας του Σαχέλ. Προσφέρουμε εξασφάλιση. Οι φίλοι στο Σαχέλ είναι πιο αποτελεσματικοί στρατιωτικά όταν γνωρίζουν ότι αν υπάρξει ένα πρόβλημα θα μπορέσουν να στραφούν στον Μπαρχάν, ιδίως στα καταδιοκτικά αεροσκάφη, για την βοήθεια. Αυτό διαπιστώνεται σε πολλές επιθέσεις που έγιναν πρόσφατα που οδήγησαν σε απώλεια ζωών για τις δυνάμεις του Σαχέλ, συχνά αργούν να στραφούν προς τον Μπαρχάν, δεν δίνουν επαρκείς πληροφορίες και άρα εμείς βέβαια μπορούμε, μάλλον εμείς δύσκολα μπορούμε να τους βοηθήσουμε αν δεν υπάρξει επαρκής ενημέρωση και γρήγορη έκκληση. Τελειώνοντας, να υπενθυμίσω ότι η δράση αυτή έχει νόημα όταν συνοδεύεται και στις άλλες διαστάσεις του. Βελτίωση της διακυβέρνησης, διπλωματικές προσπάθειες, διαβούλευση στο εσωτερικό κάθε, κάθε χώρας. Οι τέσσερις πυλώνες που καθόρισε η σύνοδος του, ΚΟ, του ΠΟ έχει ακριβώς αυτό το στόχο, να φέρει κοντά τις διάφορες προσεγγίσεις. Πρώτος, ο στρατιωτικός. Δεύτερον, ενίσχυση των εσωτερικών δυνατοτήτων της χώρας και εδώ δουλεύουμε. Και άλλοι πυλώνες που, μας που αφορούν έμεσα τον γαλλικό στρατό, αλλά που είναι σημαντική. Επιστροφή του κράτους και της διοίκησης σε όλη την περιοχή, σε όλη τη χώρα, κάτι που είναι αναγκαίο για να μπορέσουν οι περιοχές αυτές να βγουν από την κρίση τους. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, βρεθεί. Το είπατε. Οι χώρες που συμμετέχουν στι επιχειρήσεις στο Μάλι, Μπαρκάνη ιδίω, στην Μπαρκάνι ιδίω, ε, περιλαμβάνουν και την Εστονία. Θέλω να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ρέκαν για να μας πείτε ε, τη δική σας ε, άποψη για τη συμμετοχή των εστονικών δυνάμεων στη στρατηγική επιχειρήση και την θεωρήσή σας για σήμερα, ε, για την τωρινή κατάσταση και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ όπως πριν από λίγους μήνες. Ε, πρώτα απ' όλα, να πω ότι η Εστονία συμμετέχει στις διεθνείς επιχειρήσεις στην περιοχή του Σαχέλ από το 2013. Έχουμε στείλει στρατεύματα στο Μάλι από την αρχή της σύγκρουσης στο Μάλι. Η δική μας συμμετοχή στην περιοχή έχει ε, οργανωθεί σε τρεις επιχειρήσεις, τη USM και την Γαλλική Μπαρκάν ε, και την Μινούσμα. Από τις 9 Μαΐου 2018 έχουμε οργανώσει τις δυνάμεις μας και ήταν ζωτική σημασία για μας να συμμετέχουμε στην επιχείρηση Μπαρκάν και στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τις αρχές του Μάλι. Ήταν περίπλοκες, αλλά φτάσαμε σε συμφωνία. Γι' αυτό εκτιμούμε ιδιαίτερα την βοήθεια της Γαλλίας. γιατί δεν είχαμε μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τις αφρικανικές χώρες. Το 2020 η, η πρόσφατη προσφορά της Εστονίας στην επιχείρηση Μπαρκάν διπλασιάστηκε. Οι δικές μας δυνάμεις είναι έτοιμες να φύγουν από το καλοκαίρι. Και θα πάρουμε μέρος στην επιχείρηση Τακούμπα από το καλοκαίρι. Τώρα για τη συνεργασία με τους γαλλικούς υπευθύνους στην επιχείρηση Μπαρκάν, ε, οι αντιδράσεις των δικών μας στρατιωτών είναι πολύ θετικές ως τώρα. Για να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, τα στρατεύματά μας με ένα τάγμα ασχολούμαστε με την περιπολία μια συγκεκριμένη περιοχή 20 χιλιόμετρα περίπου προστασία ε, αμάχων και δύναμη κρούσης. Αυτά κάνει το δικό μας το Σύνταγμα. Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα το κλίμα και ο καιρός. Οι στρατιώτες μας που έχουν εμπειρία από το Αφγανιστάν και το Ιράκ λένε ότι ήταν πανεύκολο σε σχέση με το κλίμα του Μάλι. Φτάσανε βέβαια αρχικά Αύγουστο μήνα και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Ήδη όμως μάθαμε πώς να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις δύσκολες αντίξωες κλιματικές συνθήκες. Έπειτα είναι σαφές ότι υπάρχει και το γλωσσικό εμπόδιο. Δύσκολο να πρέπει εμείς να μιλήσουμε και να συνεννοηθούμε γαλλικά και αντιστρόφως, οι Γάλλοι να πρέπει να συνεννοηθούν στα αγγλικά μαζί μας. Μετά από 1,5 όμω χρόνο τα πάμε καλύτερα. η διαλειτουργικότητα στο κομμάτι της επικοινωνίας είναι απαραίτητη και ήδη κάτι, κάτι γίνεται. Στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν είχαμε κάποια θέματα με τις Βρετανικές δυνάμεις. Είχαμε κάποιες δυσκολίες, αλλά τα θέματα κατά κύριο λόγο επιλύθηκαν και μετά για την διοικητική μέρημνα. Την επιμελητία μέχρι τώρα Έχουμε χρησιμοποιήσει την οδό Ταλίν ε, ε, Κωνσταντινούπολη Μπαμάκο, αλλά Τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά την EMA ως καταληκτικό σημείο από το Τάλιν. Και στον ΚΑΟ. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν τη Γαλλία εδώ για την στήριξή της. και ελπίζουμε ότι η κατάσταση στην περιοχή θα βελτιωθεί τα ερχόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε και τους τέσσερις. Και τώρα να δώσω το λόγο στους βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Ντονζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Έχω πολλά να πω, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω τα εξή. Δεν υπάρχει κανένα θέατρο πολέμου όπου οι Ευρωπαίοι είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στο πλαίσιο του ΟΗΕ είτε στο επίπεδο της επιχειρήσης Μπαρκάν ή υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέατρο πολέμου που να υπάρχουν τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι που να δρούν ταυτόχρονα στρατιωτικά αλλά και οικονομικά. Το υπενθυμίζω, διότι δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν πιστεί, ε, ιδίω σε αυτή εδώ την ε, Επιτροπή, ε, για τη σημασία και την σοβαρότητα αυτής της περιοχής. Την περασμένη εβδομάδα άκουσα πολλούς στο Στρασβούργο να κάνουν ένα μπραντεφέρ και να λένε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, εξηγώντα σημαίνει στου ΔΕ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στη Μέση Ανατολή, αλλά να κρυβόμαστε και πίσω από του Αμερικάνου. Ε, και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά στο Σαχέλ ελάτε γιατί θα βρείτε χώρο να κάνετε αυτά που θέλετε. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο δυνατοί σε υπόλοιπε περιοχέ. Στην Αφρική υπάρχει χώρο για όλου. Υπάρχει πολύ πράγμα να γίνει. Ε, δεύτερο, Κρίμα που έφυγε η κυρία Ράσμουσεν. Άκουσα αυτά που είπατε, τα σημειώνω. Αλλά πρέπει να σημειώσω και λυπούμε που το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Η στρατηγική μας για το Σαχέλ έχει χαραχθεί εδώ και 9 χρόνια. 9. Το 2011 το Συμβούλιο, το Μάρτιο του 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι τα 28 κράτη, 27 τότε χωρίς την Κροατία, τα 27 κράτη είχαν υπογράψει μια στρατηγική για το Σαχέλ, που καθόριζε τα πάντα για την ε, διάρθρωση άμυνας ασφάλειας πριν, πριν τα προβλήματα με τους τζιχαντιστές που προέκυψαν το 2013. Τα είχαμε ήδη καταρτήσει όλα και 9 χρόνια μετά πρέπει να καθόμαστε να σκεφτόμαστε πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Πώς θα επινοήσουμε ξανά τον τροχό Ε, μακάρι επιτέλους κάτι να γίνει, τόσο το καλύτερο, αλλά επί εννέα χρόνια τι κάναμε. Διότι όλα τα βασικά στοιχεία για τη διάρθρωση τη ε, ασφάλεια με την ε, ανάπτυξη, για τι σχέσει με τι τοπικέ αρχέ, τα λέμε εδώ και χρόνια και δεκαετίε. Είναι κάτι που πραγματικά δημιουργεί φοβερέ απογοητεύσει, αλλά τέλο πάντων, αν μπορούμε από τώρα να κάνουμε κάτι και να προχωρήσουμε, είναι ήδη μια πρόοδο. τώρα, κάποιε παρατηρήσει για το στρατιωτικό επίπεδο. Το θυμήσατε όλοι, ξέρουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα εκεί και δυστυχώς είχαμε πολλές αυταπάτες για τις δυνατότητες των χωρών G5 του Σαχέλ. Πιστεύουμε ότι οι χώρες αυτές ήταν ε, η λύση θαύμα. Αλλά όπως το είπατε κι εσείς, ο Γάλλος Επιτελάρχης πριν από 7 χρόνια είχε αναλάβει να οδηγεί τις δυνάμεις μας στο Μάλι η γαλλική παρουσία τώρα θα πρέπει να δει τι κάνει η Ευρώπη από τη δική της πλευρά. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τις δυνάμεις στο Μάλι να ε, οργανώνουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις από κοινού. Θα πάρει πολύ καιρό για να είναι αποτελεσματική. Έχουν τεράστιες εθνικές ευαισθησίες και ευθυξίες και εδώ 105.000 5.000 χιλιόμετρα μακριά είναι πολύ εύκολο να ε, κάνουμε κρίσεις και αξιολογήσεις. Όμως, ο ανθρώπινος παράγοντος είναι πολύ διαφορετικός από τη μία χώρα στην άλλη. Τώρα τι να πω για το στρατό της Μπορκίνα Φάσο, δεν το λέω επικριτικά, αλλά η κατάσταση είναι καταστροφική. Το τι κάνουν ε, λοιπόν ε, στην Πουρκίνα Φάσο και στο Μάλι, τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά στα στρατεύματά του. Το να συνεργαστούν όλοι αυτοί μαζί και αποτελεσματικά είναι κάτι που θα πάρει ε, πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν πολύ αισιοδοξοί, ελπίζοντα ότι με λίγη χρηματοδότηση και ένα μικρό πλαίσιο θα μπορέσουν τα πέντε κράτη του Σαχέλ να δράσουν και μάλιστα αμέσω. Πρέπει αυτή την πραγματικότητα να τη δεχτούμε και θα πάρει ακόμα καιρό. Είναι λοιπόν μια πολιτική αυτή παρατήρηση και το λέω σε όλους σας, εδώ η αναπτυξιακή βοήθεια, όσο μαζική και να είναι προς τις χώρες αυτές, θα το πω κάπως ε, ανακριτολογικά, αλλά στο Μάλι ουσιαστικά ενισχύσαμε την αγορά κινήτων και τη φούσκα κινήτων στην πρωτεύουσα. Ε, στο κέντρο και για να μην πω για το βορρά της χώρας. Η αδυναμία του κράτους του Μάλι να οργανωθεί για να προσφέρει ε, πρωτογενείς υπηρεσίες στον πληθυσμό της. Εκπαίδευση, ε, υγειονομική περίθαλψη, δικαιοσύνη. Αυτό είναι ουσιαστικά ε, το σημείο που επιτρέπει να αναπτυχθεί η τρομοκρατία. Διότι δεν υπάρχουν βασικές υπηρεσίες για τους πολίτες του Μάλι, ενώ οι τρομοκράτες με τις για συνδέσεις που έχουν με τους τοπικούς με, με τις τοπικές κοινότητες μπορούν να οργανώσουν αυτά που του λείπουν από το κράτο. Οι τοπικέ αρχέ, λοιπόν, παρά τα κονδύλια που λαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Και όταν ε, του καλείται να τα κάνουν, λένε ότι είσαστε νέοι απεικιοκράτε. Έχουμε, λοιπόν, ε, μια μεγάλη πολιτική δυσκολία, η οποία δεν θα επιληθεί τώρα αμέσω. Πρέπει όμω τα κράτη δικαιούχοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν και κάποιε προποθέσει για να προσφέρουμε τη βοήθειά μα και αν δεν μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα ή δεν θέλουν να εφαρμόσουν προγράμματα διότι δεν ταιριάζουν με τη δική τους ε, πολιτική ατζέντα, ε, δεν έχουμε ε, κανένα λόγο να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να τους στηρίξουμε. Και ε, όλη αυτή η κοινή γνώμη με την νέο απεικαιοκρατία της Γαλλίας και τη Ευρώπη είναι ανυπόφορη. Ε, είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Δεν είναι και για να εξυπηρετήσουμε τα χρήματα αυτά τη Αφρικανική ελίτ των χωρών αυτών. Θέλουμε να στηρίξουμε του κατοίκου των χωρών. Αυτό που συμβαίνει στο Μάλι πραγματικά είναι ανυπόφορο. Κανένα από τι διάφορε κοινότητε στο κέντρο του Μάλι, που είναι το πιο αδύναμο σημείο τη χώρα, δεν έχει δει σχολείο, ένα κέντρο υγεία ή ένα δικαστηριάκι. Ε, και αρνούνται οι τοπικοί θύνοντες να πάνε ως εκεί. Ε, οπότε βυσοδομούν οι τζιχαντιστές με τη στρατολόγηση να ε, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται ακριβώ με τι ειρηνευτικέ συμφωνίε. Υπάρχουν υποτίθεται ειρηνικέ συμφωνίε που κανονίζουν την ανάπτυξη των στρατευμάτων και την αλληλουχία των προσπαθειών μα. Ε, ειρηνευτικέ συμφωνίε που ουσιαστικά είναι τελείω εύθραυστε από ό,τι φαίνεται. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Ε, αλλά πού ε, έχουν φτάσει τώρα, γιατί σίγουρα σταθεροποίηση του Μάλι περνάει από εκεί και μετά αισθητοτικη παρουσία. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα φύγουν από την ε, Αφρική. Αυτό είναι σαφώς ανησυχητικό, γιατί ακόμη και αυτό το ελαφρύ αποτύπωμα που αφήνουν είναι βασικά για μας. Εμείς δεν έχουμε στρατηγική αυτονομία στο συγκεκριμένο τομέα, ό,τι και αν λέμε. Χρειαζόμαστε και τη στήριξη της Αμερικής εκεί ε, για να μπορούμε να δράσουμε όπως και στο κέρας της Αφρικής. Οπότε πρέπει να δούμε σε τι, ε, με τι τρόπο και πόσο πολύ θα φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Όλεκας για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, το θέμα είναι δύσκολο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Μιλούμε για μια επταετή περίοδο. Συμμετοχή σε ένοπλων στρατιωτικών δυνάμεων. Τα νούμερα και τα μεγέθη που μας παρουσιάσατε είναι απεσιόδοξα και εντυπωσιακά. Συμμετέχουμε στο Μαλί, στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στη Σομαλία και αλλού διάφορα χρόνια. Έχουμε και τη μηνούς μας στο Μαλί. Ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος ε, πώς προσεγγίζουμε τον πληθυσμό στην αποστολή μας. Μήπως πρέπει να επανασχεδιάσουμε τις δραστηριότητε μας και να με βάση την ενοποιημένη προσέγγιση. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Επιπρόσθετη πόρη ήταν το θέμα της συζήτησης. Αυτόνομη δέσμευση ως Ευρωπαίοι. Αυτόματη εμπλοκή και αυτόνομη εμπλοκή. Τι μας προτείνεται πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πιο, ενεργά, ε, πιο ενεργά και το στρατιωτικό μας σκέλος αλλά και τον τοπικό πληθυσμό. Ίσως δεν φτάνει η εντολή. Απλά να υπάρχει μια εντολή για την Ευρωπαϊκή Αποστολή Εκπαίδευσης. Ίσως η εντολή πρέπει να διευρυνθεί. Οι φίλοι μας κάνουν ε, πολλά με τους δικούς τους συμμάχους, όμως μετά από 7 χρόνια έχουμε περισσότερες απώλειες και θύματα σε αυτή την περιφέρεια παρά ποτέ. Και έχουμε και νέες κρίσεις, όπως τις εξηγήσατε. Άρα, τελικά δεν καταφέραμε να φτιάξουμε θερμές σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό και δεν έχουμε και την ικανότητα να κατασυγάσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις. Ευχαριστώ. Για το ΡΙΝΙΟ, ο κύριος Οστρεβίσιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε να μας μιλήσετε για αυτό το τόσο επίγον ζήτημα. Δεν έχει σταματήσει να είναι επίγον το ζήτημα αυτό, άρα είναι λογικό να περιμένει κανεί να παραμείνει φλέγον ζήτημα και επίγον και τα επόμενα χρόνια. Εάν η απάντησή μα δεν είναι αποτελεσματική και δεν έρθει στην κρίσιμη και κατάλληλη χρονική συγκυρία. Πράγματι, για την ασφάλεια τη Ευρώπη οι προκλήσει είναι πολλέ. Είναι απλά θέμα χρόνου να υποστούμε αυτά τα αρνητικά και αυτούς τους κινδύνους και τις απειλές ασφάλειας με διαφορετική ίσως μορφή και διαφορετικό επίπεδο προς τον αντίκτυπο, τον αρνητικό που θα έχει στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Τι είδου απάντηση ήταν αυτή που επιφύλαξαν τα κράτη-μέλη στην περιοχή αυτή μετά τη διοργάνωση όλων αυτών των διασκέψεων και τη διοργάνωση και των μελλοντικών διασκέψεων. Αισιοδοξείτε ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη θα απαντήσουν θετικά και θα θελήσουν να συμβάλλουν στρατιωτικά, πολιτικά, ε, να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν πέρα από την απλή υπογραφή της κοινή δήλωσης ή της κοινή διακήρυξης. Τι περιμένετε. Και επίσης, αν ε, ε, σας ρωτήσει κάποιος για το τι σας λείπει περισσότερο. Έχετε λήψεις γενικές, αλλά τι σας λείπει για, τη στρατιωτική απο, απάντηση. Η ανθρώπινη πόρη ή το υλικό. Ποιο από τα δύο είναι ε, η πιο φλέγουσα ανάγκη να, ε, ανάγκη να καλυφθεί. Για το στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων ε, ενώ. Ο Αγνώ έχει απόλυτο δίκιο μίλησε για τελικά για αυτή το εγχείρημα, της, αυτή την προσπάθεια δημιουργίας κράτους. Ε, λείπουν τα βασικά. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τα αποτελέσματα, τις αλλαγές, τις οποίες να μπορεί να αντιληφθεί αν δεν υπάρχουν σχολεία, αν δεν υπάρχει βασικό ε, σύστημα υγείας, αν δεν υπάρχουν τέτοιες βασικές ε, υπηρεσίες, είναι πολύ εύκολο να έρθει κάποια ομάδα και να χειραγωγήσει τις νοοτροπίες, τον τρόπο σκέψης, την αντίληψη του, του τοπικού πληθυσμού. Πρέπει να προσανατολίσουμε τις προσπάθειές μας στην, ε, στο χτίσιμο, στην οικοδόμηση δυνατοτήτων, στο να φτιαχτεί κράτος. Και μπορούμε μετά να περιμένουμε θετικά αποτελέσματα μετά από χρόνια και ίσως και επέλθει και κάποια αλλαγή. αλλιώς, το μόνο που θα κάνουμε είναι να ε, περιστρεφόμαστε ε, γύρω-γύρω από το ίδιο σημείο και τελικά να μην καταλήγουμε πουθενά. Στα υποστηρικτικά έγγραφα διαφαίνεται πολύ χειρό το εξής μήνυμα. Δεν ξέρω γιατί έγινε ειδική μνημεία στα γαλλικά στρατεύματα, όμως μειώνεται ε, σταδιακά η αποδοχή της ξένης στρατιωτικής παρουσίας από τον τοπικό πληθυσμό. Ο, ρωτώ, ο ο τοπικό του πληθυσμός έχει θέμα με τη γαλλική παρουσία ή οποιαδήποτε ξένη παρουσία ακόμα ε, και αν αυτή λαμβάνει χώρα υπό την αιγίδα του, του ΟΗΕ των Ηνωμένων Εθνών. Ε, την αντιλαμβάνεται αρνητικά υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, την ξένη παρουσία και τη διεθνή παρουσία, γιατί αν ναι θα πρέπει να σχεδιάσουμε διαφορετικά ενδεχομένω την πολιτική μα και να την επαναπροσδιορίσουμε. Και τέλο, μπορείτε να μας περιγράψετε καλύτερα τις ε, αντιτιθέμενες δυνάμεις ποιοι είναι αυτοί που στρέφονται κατά των εθνικών στρατευμάτων και των δικών μας στρατευμάτων. Είναι ξένοι, είναι ντόπιοι. Είναι, έχουν έδρα διασυνοριακή και κινούνται μεταξύ Μαλή και Μπουρκίνα Φάσο ε, και Νίγηρα και αλλού. είναι εύκολο να περνάει κανείς σε αυτά τα σύνορα και να πολεμάει δεξιά και αριστερά και άρα να αναπτύσσεται σε περιφερειακή δύναμη. Ε, είναι άνθρωποι που βασίζονται σε φυλές και ολόκληρες φυλές έχουν προσχωρήσει σε αυτές τις ε, τάξεις. Ποιοι ακριβώς είναι και πώς, επιδεινώνεται η κατάσταση ασφαλείας ε, και πώς θα επιδεινωθεί περισσότερο με την αποκαλούμενη μεταναστευτική κρίση. Δηλαδή αυτοί που μας πολεμούν και που στρέφονται ενάντια στον τοπικό πληθυσμό. Είναι οι ίδιοι που εμπλέκονται ως διακινητές ε, και που προσπαθούν να στείλουν ε, μετανάστες στην Ευρώπη και έτσι να έχουν ε, πολύ μεγάλο πλούτο από αυτή την πηγή και να έχουν μια πηγή χρηματοδότηση πολύ σημαντική. Πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα τις απαντήσεις σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασέσκου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Ε, τα αγγλικά μου ενδεχομένω δεν είναι πολύ καλά. Τα ρουμανικά είναι τα καλύτερα. Και νομίζω ότι είναι καλύτερα να με ακούσετε στα ρουμανικά παρά στα αγγλικά ή και ακόμα χειρότερα θα ήταν στα γαλλικά. Ήθελα λοιπόν να σας, να σας πω τα εξής. Ως προς την προετοιμασία της αποστολής έχουν διατυπωθεί διάφορες επικρίσεις αλλά και οι αντιδράσεις των δικαιούχων κρατών είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή η έκθεση τα απεικονίζει αυτά με πολύ αρνητικά χρώματα. Ε, τελικά χάνουμε το χρόνο μας με ορισμένους ε, εταίρους. όλα αυτά τα γράφει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ή τέλο πάντων ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κανείς εύκολα ε, διαβάζοντας την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Τι κάνουμε λοιπόν όταν ο δικαιούχος των αποστολών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά δεν θέλει αυτή τη στήριξη. Σπαταλούμε χρήματα και στρατιωτική προσπάθεια. Και οι δικαιούχοι τελικά δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Έτσι κατανοώ και έτσι ανταλαμβάνομαι την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να λαμβάνει η χώρα ε, μια παρέμβαση σε πολιτικό επίπεδο να διευκρινίσουμε τι θέλουν οι δικαιούχοι της δικής μας παρέμβασης. Η περιοχή του Σαχέλ είναι τεράστια. Εκτείνεται σε μια απέραντη γεωγραφική έκταση. Το είπε και ο αντιστράτηγος. Δεν μπορεί κανείς να ε, επιβάλλει λύσεις στρατιωτικές εκεί με 4.500 στρατέματα μόνο. Σε μια απέραντη έκταση. Αν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, τότε πρέπει πραγματικά να λυπόμαστε τις φορές που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την απόψή μας, αλλά και να δουλεύουμε για να καλλιεργήσουμε την αλληλεγγύη στην περιοχή αυτή. Η Γαλλία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος όλων αυτών. Μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστορία για να αντλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα Ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν πιο ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία και κατά επέκταση να εμπλακούν και να συμμετάσχουν περισσότερο σε αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στον, στους Ευρωπαίους, γιατί αυτή η επιχείρηση στο Σαχέλ φαίνεται να μην τελειώνει ποτέ. Είναι σαν πηγάδι χωρίς ε, πάτο, στο οποίο να ρίχνουμε συνεχώς χρήματα, να βάζουμε χρήματα τα οποία να χάνονται και τελικά να μην καταλήγουμε σε κανένα αποτέλεσμα. Και όλα αυτά συνεπάγονται επίσης μια τεράστια διπλωματική προσπάθεια. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε καλούς εταίρους, ε, αυτοί που δικαιούνται τη στήριξή μας να γίνουν καλή εταίρημο, μας και να έχουμε και σωστό εξοπλισμό, επαρκή εξοπλισμό στρατιωτικό και επαρκή ε, συμμετοχή από όλα τα κράτη. Είναι μια αποστολή εμβληματική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Μετά τα γεγονότα στο Βερολίνο, ε, Παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις για την επιχείρηση Σοφία και τη Μεσόγειο. Δεν φαίνεται να θέλουμε πραγματικά να εμπλακούμε και να είμαστε παρόντες στο ΣΕΧΕΛ. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διπλωματική προσπάθεια από μόνη της δεν φτάνει. Όπως βλέπετε, με τις πρόσφατες εξελίξεις χρειάζονται διπλωματικές προσπάθειες αλλά χρειάζεται παράλληλα να υπάρχει και η ικανότητα να επιβάλλει κανείς αυτό το οποίο θέλει. Για παράδειγμα, υπάρχει επίκριση προς την Τουρκία σαφέστατη όμως η Τουρκία τελικά καταφέρνει να υιοθετεί την προσέγγιση της ε, προσφεύγοντα και ε, στη στρατιωτική δράση. 4.500 στρατιώτες δεν είναι αρκετοί λοιπόν για το Σαχέλ και η, μια περιορισμένη αποστολή με ε, εντολή πολύ περιορισμένη δεν φτάνει. Θα έπρεπε να είναι πιο διευρυμένη η εντολή. Νομίζω ότι πρέπει σε βάθος όλη αυτή η παρουσία μας εκεί να αναδιαρθρωθεί, να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων και να ε, συνομιλήσουμε με το στρατιωτικό προσωπικό ε, έτσι ώστε με τη βοήθειά του να καταλήξουμε στην ε, καλύτερη δυνατή εντολή. Δεν είμαι εμπειρογνώμας, δεν είμαι ειδήμων ούτε ειδικό για την κατάσταση αυτή. Αν διαβάζω, διαβάζοντας όμως την ε, έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, καταλήγω ε, σε αυτά τα συμπεράσματα. Και νομίζω ότι όποιος τη διαβάσει προσεκτικά την έκθεση αυτή θα καταλάβει ότι η έκθεση ουσιαστικά λέει ότι σπαταλούμε χρήματα. Άρα τίθεται το ερώτημα, πόσα περισσότερα χρήματα θέλουμε να σπαταλήσουμε ή για πόσες περισσότερες δεκαετίες. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, είναι σαφέστατο ότι δεν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά διατηρούμε ένα status quo, το οποίο δεν ωφελεί ούτε τα κράτη στην περιοχή του Σαχέλ, ούτε μας ευνοεί εμάς και μας βολεύει σε τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το... Δίνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους ομιλητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν καταλαβαίνω τη σημασία αυτών που έκαναν σε αυτό το σημαντικό τομέα, αντιλαμβάνομαι και τους κινδύνους που διατρέχουν. Η ερώτηση μου είναι εξή. Την περσμένη εβδομάδα εγκρίναμε στο Στασβούργο μια έκθεση για την εφαρμογή της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Έκθεση του συναδέλφου κ. Ντανζόν. Έχω την εξή ερώτηση για την έκθεση αυτή. Τι λέτε εσείς για το σημείο 35 της έκθεσης. Για να σας βοηθήσω με την απάντηση, θα διαβάσω τι αποφασίσαμε, τι εγκρίναμε στο Στρασβούργο. Και λέω, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν ανέφερε ιδιαίτερους δείκτες παρακολούθησης των ε, αποτελεσμάτων στις αποστολές στον Ήγηρα και το Μάλι, ενώ η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ε, αυτών ήταν ανεπαρκής και δεν λήφθηκε επαρκώς υπόψη οι συνέπειες που θα είχαν. Η ερώτηση μου είναι, εσείς τι άποψη έχετε για αυτό το σημαντικό σημείο που εγκρίναμε στο Στρασβούργο την περσμένη εβδομάδα. Κύριος Γουάλλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Σκοτεινή εικόνα που δώσατε. Έχω την εντύπωση ότι παρά την στρατηγική που ακολουθούμε εδώ και χρόνια, τα πράγματα δεν βελτιώνονται. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνεται. Ο, Αϊνστάιν είχε πει στο παρελθόν ότι όταν κάνουμε τα ίδια πράγματα και περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα είναι μια μορφή παράνοιας. Πιστεύετε ότι είναι δυνατή μια στρατιωτική λύση ή πιστεύετε ότι χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση. Αν κατάλαβα σωστά, συμφωνείτε ότι τα κράτη εκεί είναι τόσο τροτά και ευάλωτα που συνιστούν λείπασμα για την ανάπτυξη τζιχαντιστικών δυνάμεων. Αν η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπιστεί, αν δηλαδή δεν αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, το επίπεδο φτώχεια στην περιοχή και δεν το βελτιώσουμε, θα παραμείνει η κατάσταση πολύ δύσκολα για να επιτευχθεί μια στρατιωτική λύση. Πολλές οι ερωτήσεις που σας τέθηκαν. Να σταθώ και, εγώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, ιδίω ως προς το τι λείπει στην αποστολή για το Μάλι, ούτω ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Είναι θέμα προσωπικού, είναι θέμα εντολής, είναι θέμα δυνατοτήτων, παροχής δηλαδή δυνάμεων και εξοπλισμού ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να έχει στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη π.χ. Επίσης, υπήρξαν κάποια ευρωπαϊκά κράτη που έδειξαν ενδιαφέρον να μετάσχουν. Φερρυπίν στο πλαίσιο της επιχείρησης Τακούμπα Έχουμε κάποια καλύτερη εικόνα για τα κράτη που ανταποκρίθηκαν θετικά. Άλλοι πολλοί ομιλητές ε, σχολίασαν το ρόλο των εξωτερικών εταίρων, εξωτερικών και στη ζώνη και στην Ένωση. Ποιος μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο. Η ομάδα των 5 για το ΣΕΧΕΛ έχει μια κριτική δεν θα έλεγα, τέλο πάντων διαυγή αντιμετώπιση του τι του ζητούμε. Τηρήθηκαν οι υποσχέσεις ωστόσο. Τι γίνεται επί τόπου ως προς την παρουσία άλλων δυνάμεων με άλλες προτεραιότητες σε σχέση με εμάς. Η κυρία Μάρκουσον πρώτα και μετά οι υπόλοιποι όπως θέλουν. Η κυρία Μάρκουσον. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Πολύ καλές οι ερωτήσεις. Ξεκινώ με την ερώτηση για το ότι είχαμε μια στρατηγική από το 11 που βρισκόμαστε σε φάση αναθεώρησης. Η συζήτηση μαζί σας αυτό το στόχο έχει μεταξύ άλλων. Δύο μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν και που συζητούμε με την ομάδα των πέντε είναι ότι χρειάζεται να καταλάβουν αυτή την κρίση. Κάποιος αναφέρθηκε στην ειρηνευτική διαδικασία στο Μάλι. Πολύ καιρό δίναμε έμφαση στο Μάλι. Τώρα έχουμε επιθέσει τον Μπουρκίνα Φάσο, στο Νίγηρα, στο Τσάντ, με άλλα προβλήματα, στη Μαυριτανία. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Μπορώ να σας πω ότι σε πολλές ευκαιρίες είχα πάει με την ύπα του εκπρόσωπο σε πάρα πολλές συναντήσεις όπου καταστήσαμε σαφές πως οι κυβερνήσεις των χωρών πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Και αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Εντοπίσαμε μαζί τους ειδικέ έφορες ζώνες τις λέμε, όπου αν δείτε την ιστορία του Σαχέλ, πάντα υπήρχαν τεράστιες περιοχές νομαδικής κατοικίας. Πολλές, δηλαδή η έμφαση που δόθηκε από τις δημοκρατικές οργανώσεις είναι εκεί που δεν υπήρχε μεγάλη παρουσία του κράτους ποτέ. Άρα εμείς θέλουμε να συνδέσουμε την ασφάλεια με την ανάπτυξη. Για να απαντήσω στο ερώτημα αν η ασφάλεια περνάει μόνο. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί τη μία μέρα είναι κανονικοί πολίτες, την άλλη μπαίνουν στο λαθρεμπόριο ή στο αντάρτικο. Είναι και η λογική των περιοχών αυτών. Πολλά είναι τα θέματα που μπορεί να σχολιαστούν για το θέσιμο. αυτό, ίσως και ο στρατηγός να τα πει. Αυτό που θέλουμε να και συζητούμε τώρα είναι μεταρρυθμίσεις. Υποστήριξη στις μεταρρυθμίσεις, υποστήριξη στην κυβέρνηση για να ασκήσει μεταρρυθμίσεις και εντοπισμός των γεωγραφικών περιοχών που χρειάζεται η παρέμβαση από μας και ανθρωπιστικά και στρατιωτικά και πολιτικά, προσφέροντας στους ανθρώπους των περιοχών αυτών εναλλακτικέ κανονικής διαβίωσης. Υπήρχε μια ερώτηση για την ελευθερική διαδικασία στο Μάλι. Ήμουν στην τελευταία συνάντηση στις 19 του μηνός, ε, προχτές, όπου αναγγέλθηκε πως η συνάντηση θα ήταν ιστορική, γιατί δεν είχαν συναντηθεί για πέντε μήνες, λόγω του θέματος του Τιντάλη. Οι Νιγηριανοί είναι εκεί τώρα με τον Υπουργό τους. Ήρθε και η Αλγερία, πέντε υπουργοί του Μάλι μετήχαν, θα γίνει μια αναδίπλωση στο θέμα του Τιντάλ και θα ενισχυθούν πολιτικές ανάπτυξης με πόρους που θα είναι στραμμένοι κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας. Τώρα, να επανέλθω στην αναθεώρηση της στρατηγικής. Αυτό είναι βασική μας προτεραιότητα και οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ, οι απόψεις οι δικές σας απόψεις που ακούμε βοηθούν πολύ. Μετανάστευση, το τελευταίο θέμα. Ήμουν παλιότερα πρέσβης της Δανίας, στον Μπουρκίνα Φάσο και στον Ήγηρα, στο παρελθόν. Πολλά πράγματα στην περιοχή αυτά, αυτή συνδέονται μεταξύ τους. Το μεταναστευτικό συνδέεται και με τον παράνομο τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κάνει τη ζωή του. Υπάρχουν αυτοί, αυτές οι παράνομες διαδρομές, οι διαδρομές δηλαδή μεταφοράς παρών παράνομων που τη μία μέρα μεταφέρουν ανθρώπους τα όπλα, την άλλη μέρα όπλα. Πρέπει να συνεργαστούμε με το, συνεργαζόμαστε με το Μάλι και με την Αφρικανική Ένωση για ένα παρατηρητήριο στο Μάλι που θα μας δώσει περισσότερη γνώση για τις διαδρομές της μετανάστευσης στην Αφρική. Το θέμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη βέβαια συζήτηση, αλλά ε, είναι κρίσιμο και αυτό το θέμα. Σύνθετη λοιπόν η διαδικασία, σύνθετα τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο στρατηγός. για να απαντήσω για την, για Αμερικανική εμπλοκή. Η κατάσταση μετά την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας η εμπειρία και η γνώση που έχουν αποκτήσει για μας οι αντίπαλοι μας, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο την αμερικανική υποστήριξη. Σε όλη την Αφρική, όχι μόνο εκεί. Έχω ταξιδέψει, θα πάω την Κυριακή στη ΣΥΠΑ και ένα από τα μηνύματα που θα τους πω είναι μην ξεχνάτε την Αφρική. Είναι θέμα διατλαντικής ασφάλειας, όχι ευρωπαϊκής, αλλά αυτό πρέπει να το πούμε το συντομότερο δυνατό. για τις αποστολές e UTM. Εξετάζουμε προφανώς το πώς, πού θα οδηγήσει η αύξηση των ξένων μαχητών στο Σαχέλ. Έχουμε ήδη κάποια δακτυλικά αποτυπώματα. Μαθαίνουν γρήγορα οι αντίπαλοι αλλάζουν τις τακτικές, τις τακτικές τους, αλλάζουν τις διαδικασίες και μαθαίνουν από τα λάθη που έκαναν στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των επιτόπιων δυνάμεων. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τους εξαιρετικά ευφύης και επινοητικούς τζιχαντιστές. Επίσης, η τοπική κατάσταση είναι προβληματική. Υπάρχει μια μεγάλη ματέωση των νέων που δεν βρίσκουν δουλειά και που είναι έφορο έδαφος για προσιλητισμό από τους τσιχαντιστές. Έτσι ξεκίνησε και η ISIS στη Συρία και στο Ιράκ. Ε, απευθυνόταν σε νέους κάνοντάς τους τζιχαντιστές. Η ίδια λογική ακολουθείται και εκεί και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Για την αποστολή στο Μάλι και τις προοπτικές της. Συμφωνώ μαζί σας ότι και εμεί είμαστε απογοητευμένοι που τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που προσδοκούσαμε, δεν είναι αποτελεσματικά, δεν έδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα σε 7-8 χρόνια εκεί χωρίς αλλαγές. Βεβαίω έχει αλλάξει η κατάσταση. Είναι άλλα τα, τα προβλήματα τώρα, άλλα πριν από 3-4 χρόνια. Άλλα διακυβεύονται τότε, άλλα τώρα. Βέβαια, κάναμε πράγματα. Είναι μια πολύ καλή επένδυση η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει υψηλή. Οι εκπαιδευτές μας είναι πάντα ευπρόζεκτοι, δεν έχουμε διαδηλώσει εναντίον μας. Διαφορετικό βέβαια το θέμα είναι το πώς εμπλεκόμαστε στρατηγικά στη μάχη και τι γίνεται αυτό, αλλά ε, δεν έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει αντι, εχθρική αντιμετώπιση. Τώρα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της Ένωσης για να έχουμε μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση. Η απάντησή μου είναι στρατιωτική λύση δεν υπάρχει μόνο στρατιωτική λύση. Ούτε στη δική Αφρική, ούτε παντού. Η δύναμή μας είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε στρατιωτικές δραστηριότητες της Ένωσης και άλλες δραστηριότητες της Ένωσης αφού έχουμε τη δυνατότητα. Η εντολή που έχουμε είναι παρκής, αρκεί να επεκτείνουμε την υποστήριξή μας λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο στενά σε άλλους τομείς. Και αυτό ίσως είναι ο τρόπος για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας δεδομένου ότι έχουμε ανθρώπινους πόρους και την υποστήριξη των κρατών μελών. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δυνατότητα της Ένωσης έχει ε, βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την παροχή ε, εξοπλισμού και υποδομών, καθιστώντας την παρουσία μας λίγο πιο εύκολη. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι εύκολο για να συμπεριλάβουμε στην πολιτική μας όλες τις διαστάσεις της λειτουργίας της ομάδας των πέντε πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη να δεχθούν την υποστήριξή μας και νομικά αλλά και πολιτικά κυρίως. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι μια χώρα που θα χρειαστεί και διμερή υποστήριξη. Μελετούμε πώς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την ε, αποστολή της υποστήριξής μας εκεί, την υποστήριξη της αποστολής μας εκεί. Αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ στα να Κανένα πρόσθετο σχόλιο για την Τακούμπα, ας πούμε. Μιλήσαμε για ανάγκες και πώς πρέπει να εξελιχθούν ε, και να εκτεπλεθούν οι δυνάμεις στην Τακούμπα. Δύο στοιχεία θέλω να σχολιάσω κι εγώ. Οι γαλλικέ δυνάμεις δεν έγιναν ε, θετικά δεκτέ από τον πληθυσμό στι χώρες του Σαχέλ, υπόθηκε. Να το διορθώσω. Διότι επί τόπου έχουμε δυνάμει. Την επιχείρηση Μπαρκάν και σίγουρα ε, οι πολίτες τους δέχονται θετικά. περιμένουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ε, και τις γαλλικές οι πολίτες γιατί τους προσφέρουν ασφάλεια. και με tweets στην Παμάκο ας πούμε και με το πώς αντικατοπτρίστηκε αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά δεν είναι όλος ο πληθυσμός του Μάλι νέος. Εάν δούμε όμω ότι άλλοι έχουν διαφορετικέ πολιτικέ προτεραιότητε, το ίδιο και τα μέσα μαζική ενημέρωση, διαμορφώνεται η εικόνα αυτή ανάλογα με την πραγματικότητα. Όμω σίγουρα κάτι προσφέρουμε ε, για τον πληθυσμό στον οποίο παρέχουμε προστασία και γι' αυτό έχουμε κληθεί ω εκεί. Τώρα, η αιμονή ε, και η καρτερικότητα είναι θέμα σοφία και όχι. Και κάποιες, αλλά κάποιε φορέ μέχρι και τρέλα. Ε, η μάχη κατά του τζιχαντισμού, λοιπόν, είναι ένα αγώνα που θα κρατήσει πολύ. Ξεπερνά τι πολιτικέ βλέψει, ξεπερνά το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Θα χρειαστούν χρόνια για να σταθεροποιηθεί η περιοχή. Θα πρέπει να πολεμήσουμε την τζιχαντιστική τρομοκρατία διεθνώ και αυτό θα χρειαστεί πολύ καιρό. Χρειάζεται λοιπόν μια μακρόπνοη προσπάθεια και χρειάζεται μια σφαιρική ε, προσπάθεια πολλών κρατών και στο στρατιωτικό σκέλος. Τώρα, για το τι μπορεί να γίνει με μια ενδεχόμενη υποχώρηση των Αμερικανών και τις ανάγκες που συνδέονται με την πρόοδο των τρομοκρατών. Είναι σαφές ότι όλη η καλή αισθητοτική θέληση ε, εμάς μας βοηθάει. Στο Σαχέλ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων, δυνατοτήτων δράσης δηλαδή, και ανάλογα με τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, δημοκρατικών αποφάσεων, ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε στρατού, υπάρχει δυνατότητα να ε, λάβει κανείς μέρος στην Παρκάν προκειμένου να κάνει κάποια κίνηση κατά των τρομοκρατών, όπως λέμε εμείς ε, στη δική μας διοργάνωση, στην επιμελητεία. Ε, αερομεταφορές, μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευση, δέσμευση ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για τι ευρωπαϊκέ δυνάμει που μπορούν να εκτεπλωθούν στο Μάλι και γενικώ στο Σαχέλ. Τώρα, η συμμαχία μα για το Σαχέλ θέλουμε να αναπτυχθεί. Είναι γι' αυτό σημαντικό να μπορούμε να συνδυάσουμε τι δυνάμεις διαφορετικών χωρών σε διαφορετικά επίπεδα και ανάλογα με τι δυνατότητε του. Εάν λοιπόν φοβάστε μήπως βραχείτε ή δεν μιλάτε γαλλικά, ε, δεν υπάρχει θέμα. Ε, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σας εντάξουμε στη δύναμή μας, όπως είπε και ο στενός συνάδελφος. Και βεβαίως και στις ειδικές δυνάμεις υπάρχει χώρος, ε, με την δόνα μικρή στα κούμπα που πρόκειται να ξενολειτουργεί, ειδικό στάτευμα. Εάν υπάρξουν ευρωπαϊκές χώρες που θα ανταποκριθούν σε αυτή την έκκληση θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας για την καταπολέμηση των δημοκρατών σε αυτήν την περίοδο, περιοχή, κυρίως στο ε, και στα σύνορα Νίγηρα, Μπουρκίνα σφάσω και Μάλι. Η ειδική δύναμη Τάκουμπα θα κάνει αυτό που γινόταν ως τώρα, στο Αφγανιστάν και σε άλλα θέατρα πολεμικών επιχειρήσεων θα κοιτάζουν ε, να βελτιώσουν το επίπεδο των ε, δυνάμεων του Μάλι για να μπορούν να βγουν από ένα στρατόπεδο και να πάνε να χτυπήσουν τρομοκράτες εφόσον χρειαστούν και εφόσον έχουν ανοιχνευτεί από τα μέσα που θα έχουν συγκεντρώσει. Για τα μέσα τα ίδια, για τους ενδεχόμενους φίλους μας, γιατί ε, αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο που δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω, αλλά αν οι Αμερικανοί φύγουν, θα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο ευρωπαϊκέ δυνάμει. Θα χρειαζόμαστε αεροσκάφη, βομβαρδιστικά. Ε, θα χρειαζόμαστε εκπαίδευση με μια επανδρομένα αεροσκάφη ε, και πολλά άλλα. Οι ευρωπαϊκέ δυνάμει λοιπόν θα πρέπει. να μπορούν να υποστηρίξουν συντονισμένα το τι συμβαίνει. Σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων, λοιπόν, οι στρατιωτικές κινήσεις απαιτούν περισσότερη στήριξη. Τώρα για, την... για τα μέσα που χρειαζόμαστε. Είναι ανθρώπινα μόνο. Ρωτήσατε, όχι μόνο. Ε, είναι ένα σύνολο. Ε, και εμείς, οι δυτικές δυνάμεις, αλλά και αυτές του Σαχέλ, για να είμαστε ε, δραστικοί απέναντι σε έναν περίπλοκο και απρόβλεπτο εχθρό, Χρειαζόμαστε κόσμο, στρατιώτε, γυναίκε και άντρε, που να έχουν εκπαιδευτεί, ε, καταρτιστεί, να έχουν κινητρό, να έχουν εξοπλισμό και όπλα, να έχουν αρχηγού επικεφαλής που και αυτοί να είναι ε, ε, εκπαιδευμένοι, να γνωρίζουν τι κάνουν, να έχουν μια σαφή εντολή και να μπορούν να του οδηγήσουν να εκτελέσουν κάποια δράση, όχι απλώ να βγαίνουν μια, από ένα εδώ με την πρώτη επίθεση και να μην ξέρουν τι να κάνουν απέναντι στον εχθρό. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη αυτοπεποίθηση που περνά από εξοπλισμό, υλικό δηλαδή και εκπαίδευση, ε, κατάρτιση, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση που λείπει. Είναι θέμα και ανθρωπίνων πόρων. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν ε, κάνει ένα στρατό ε, ποιοτικό. Αυτό θέλουμε στο γαλλικό στρατό και αυτό ελπίζουμε να συμβεί αύριο και με τις δυνάμεις του Σαχέλ. Ευχαριστούμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ρεκάνεν. Αν θέλετε σύντομα, γιατί θα ολοκληρωθεί αυτό το μέρος της συζήτησής μας τώρα. Ναι. Απλώς να σχολιάσω ότι όπως λέτε Γαλλία, Βέλγιο και Ισπανία και όταν στα τέλη του 2017 ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το αν η Εστονία θα πάρει μέρος στην επιχείρηση Μπαρκάν τα ευρωπαϊκά κράτη ενδιαφέρονταν κυρίως για το στρατιωτικό σκέλος. Εμείς μοιραστήκαμε όλες τις πληροφορίες που είχαμε για την νομική διάσταση, πώς μπορεί να λυθούν, πρέπει κανείς να το λύσει διμερώς παρά το πλαίσιο του ΙΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις χώρες του Σαχέλ βασιστήκαμε στην εμπειρία που είχαμε στον τομέα αυτό από το παρελθόν και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της ευρωπαϊκής συμμετοχής στην επιχείρηση Μπαρκάν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντανζάν θέλει ένα τελευταίο σχόλιο για την κατάσταση του Μπουρκίνα Φάσου. Ναι, Πρόεδρε, απλώς να ευχαριστήσω και να τονίσω ότι αυτό που κάνει η Εστονία είναι πραγματικά αξιέπαινο. Είναι μια ευρωπαϊκή πραγματικά κίνηση. Ο καθένα καταλαβαίνει ότι η προτεραιότητα τη ασφάλεια και τη προστασία τη Εστονία δεν είναι η περιοχή του Σαχέλ. Το καταλαβαίνει και το καταλαβαίνει καθένα. Ωστόσο, η Εστονία συμμετέχει, συμμετέχει και μάλιστα αρκετά σημαντικά ω προ αναλογικά ω προ τα στρατεύματά τη. Η Εστονία έχει κατανοήσει ότι δεν μπορούμε από τη μια να απαιτούμε την αλληλεγγύη των συμμάχων για να ε, προστατεύει τα συμφέροντά μα, χωρί να μοιραζόμαστε τι ευθύνε σε άλλε περιοχέ που είναι σημαντικέ για του συμμάχου μα. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι πραγματικά αξιοσημείωτο αυτό που κάνει η Εστονία, είναι αξιέπαινο και είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ε, και παράδειγμα. Τώρα, για τις επιχειρήσεις, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, εκπαίδευσης. UTM για αυτό που είπατε και για το Μάλι. Υποτίθεται ότι πρόβλημα είναι η γλώσσα, είναι ένας φραγμός. Είναι μια χώρα γαλλόφωνη και πολλοί στατοί δεν έχουν Γάλλους αξιωματικούς να στείλουν. Γαλλόφωνους μάλλον αξιωματικούς να στείλουν. Το ακούμε συχνά αυτό το επιχείρημα. Ε, φαίνεται να στέκει, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ επέστρεψα από τη Σομαλία, όπου είχαμε μια παρόμοια αποστολή ε, εκπαιδευτική. Μόνο 7 χώρες όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση της Σομαλία, ενώ η βασική και επίσημη γλώσσα εκεί είναι τα αγγλικά. Άρα, ε, ο γλωσσικός φραγμός για να πάει κανείς στο Μάλι είναι ε, ψευδοεπιχείρημα. Ε, είναι κύβδηλο. Εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν χρειάζεται για να επιδείξει κανεί τη το του να ασχολείται με γλωσσικού φραγμού. Το αποδεικνύει το Μάλι. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω του ε, ομιλητέ μα για τι πολύ ενδιαφέρουσε εισηγήσει του σήμερα το πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω όσου από εσά θα φύγουν τώρα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα λεπτό για να περάσουμε στο δεύτερο μέρο τη σημερινή συνεδρίαση για την κατάσταση ασφάλεια στην Πορκίνα Φάσου. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αντιστράτηγο Έσα Πούλκιτσεν και την κυρία Μάρκουσεν που παραμένουν στο πλάι μας, ε, παραμένουν δίπλα μας. Θα ακούσουμε μέσω Skype τον κύριο ε, Λέμποβιτς, προσκεκλημένο ερευνητή εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξωτερικές υποθέσεις και θα μας μιλήσει και εκείνος για την Μπουρκίνα Φάσο, μια χώρα στην οποία η ασφάλεια έχει ε, χειροτερεύσει την ε, τελευταία περίοδο. Θα θυμόμαστε εκείνη τη βραδιά, χθες, 30 πολίτες βρήκαν το θάνατο, ήταν ε, άλλη μια ε, περίπτωση βίας. Έχουν γίνει τέτοια και στο παρελθόν και έχουμε και καταστάσεις εκφοβισμού των μαθητών, των δασκάλων σε διάφορα χωριά στην Μπουρκίνα Φάσο όπου διστάζουν να πάνε στο σχολείο, ο τοπικός πληθυσμός διστάζει να στείλει τα παιδιά του. Υπάρχει δηλαδή μια συστηματική επιχείρηση αποσταθεροποίησης της χώρας. Αυτές οι ταραχές στο Μαλί έχουν διαδοθεί και έχουν επεκταθεί μέχρι και την Μπουρκίνα Φάσο και αυτή η επιμόλυνση, αν θέλετε, η διάχυση των αρνητικών αυτών συνοπιών γίνεται με όλο και πιο εντατικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε παρόντες εδώ και πολλά χρόνια και ε, Είμαστε παρόντες σε τομεί που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση, με τη γεωργία, με το νερό, με την απασχόληση, με την ενέργεια, με τις δημόσιες υπηρεσίες, με την ε, αγροδιατροφική και επισητιστική ασφάλεια, μεταξύ άλλων. Πάρα πολλά χρήματα έχουν δοθεί από τα διάφορα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αρχές της χώρας αυτής δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αυτό το ξέσπασμα βίας και αυτό τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών βίας. Κύριε Λέμποβιτς, αν είστε κοντά μας στην άλλη άκρη της γραμμής, μέσω Skype, αν λειτουργεί η σύνδεση και μας ακούτε, θα σας ζητήσω να πάρετε το λόγο ευθύ αμέσω για να μας μιλήσετε ε, για τις πηγές, για, τη, ε, για τις αιστείες ε, προέλευσης όλης αυτής της αναζωπήρωσης της βίας. Από πού προέκυψε και πώς και να μας μιλήσετε για τις μελλοντικέ προοπτικές, τι μέλη με τη χώρα αυτή για την οποία η φετινή χρονιά το 2020 είναι και μια εκλογική χρονιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνετε να ε, σας μιλήσω. Πολύ λυπάμαι που δεν μπορεί ε, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας στις Βρυξέλλες. Είναι αργά το βράδυ στη Νέα Υόρκη και έχω μείνει για να ε, σας μιλήσω. Όντως είναι πολύ επικίνδυνη η κυρία αυτή στην Μπουρκίνα Φάσο ε, ε, είχαμε και άλλη μια σφαγή αμάχου πληθυσμού στην επαρχία Σαν Ματέγκα. Έχουμε 48 ώρες δημόσιο επίσημο πένθος. Το, στα τέλη του 2019 μπορούμε να πούμε ότι είχαμε περίπου ε, από 1.000 μέχρι 2.200 θανάτους. Στην Μπουρκίνα Φάσο εκατοντάδες στρατιώτες βρήκαν το θάνατο. Ε, κάθε φορά πρόκειται για δολοφονία και για άσκηση βίας. Η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα αυτή έχει επιδεινωθεί από την εισβολή των ομάδων τζιχαντιστών. Είχαμε επιθέσεις και το 16 και το 2017. Η ανασφάλεια αυτή οφείλεται εν μέρη στην πτώση του καθεστώτος Μπλέζ Κομπαορέ. Υπήρξαν εντάσεις, υπήρξαν κίνδυνοι, αλλά δεν ξεκίνησαν όλα αυτά με την αποχώρηση του Μπλέζ Κομπαορέ. Οι τζιχαντιστές έχουν καταλάβει το Βόρειο Μαλί από το 2012, η Αλκάιντα έχει προχωρήσει και τα διάφορα άλλα κινήματα τα τζιχαντιστικά στη Δυτική Αφρική έχουν εκπαιδεύσει τέτοιους μαχητές στη Μπουρκίνα Φάσα και ορισμένοι ήταν παρόντες όταν ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις ε, εναντίον του Μπλέσκο Παορέ. Και έτσι μπόρεσαν να καταλάβουν αυτό το κενό Υπάρχει ο Ιμπραχή Μαλαντίκο, θρησκευτικό ηγέτης, έχει ε, στενούς δεσμούς με τον Αχμεντίν Κούφα και έχει περάσει πολύ χρόνο στο Μαλί, έχει ε, μπει και φυλακή άλλωστε. Όταν πέθανε ο Αχμέντι το 2017, ε, τα ενία πήρε ο αδερφός του Τζαφάρ και αυξήθηκαν οι επιθέσεις. Και έχουμε τις δύο βασικές τσιχαντιστικές ομάδες την Αλκάιντα και το Ισλαμικό ε, κράτος στη Σαχάρα. Τα μέλη προσχωρούν στο EIGS. Έγιναν επιθέσεις τον Αύγουστο του 2019. Το Ισλαμικό κράτος ε, διεκδίκησε την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις και είχαμε και ε, συμμετοχή των μαχητών τσιενμάι, Είχαμε επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού, έγιναν πολλές περιπολίες. Υπάρχει κίνδυνος διάδοσης ε, αυτού του προβλήματος και στις παράκτιες χώρες της Δυτικής Αφρικής, γιατί προσπαθούν όλοι να έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Έχουμε στρατιωτικές ομάδες και ε, τοπική πολιτοφυλακή που αποτελεί το αντικείμενο των στόχων και όλο ε, και περισσότερους χριστιανούς. Αυτές οι επιθέσεις έχουν στόχο να υπονομεύσουν την αντιπολίτευση στην ομάδα και να αποδυναμώσουν την παρουσία του κράτους. Έχουν επίσης το στόχο να στοχεύσουν ε, ανθρώπους για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι πληροφορούν για την ύπαρξη ομάδων τζιχαντιστών, είναι πληροφοριδότες των γαλλικών δυνάμεων ή της κυβέρνησης της Μπουρκίναμπε. Τελικά οι τζιχαντιστικές ομάδες έχουν κεφαλοποιήσει σε πάνω σε όλες αυτές τις ε, ε, βίες πράξεις εναντίον των πολιτών οι οποίες προέρχονται από τις δυνάμεις ασφαλείας του Μπορκιναμπέ και έχουν αξιοποιήσει δηλαδή αυτή τη δυσαρέσκεια ε, αυτές, ε, αυτά τα αντίπεινα έχουν ως στόχο τις κοινότητες Φουλάνη που έχουν ε, κάτι το οποίο οδηγεί σε αυξημένο φόβο στην Μπουρκίνα Φάσο και στο Μάλι και στον Νίγηρα ε, για το ότι θα υπάρξει ξέσπασμα κινήματος τζιχάντε τύπου Φουλάνη. Όλες όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ενδεχομένως είναι υπερβολικοί και υπάρχει ο, ο κίνδυνος να ολόκληρες κοινότητες να φέρουν στίγμα ενώ ε, μπορεί να μην ισχύει αυτό. Είναι αληθές ότι οι τζιχαντιστικέ ομάδε τονίζουν ιδιαίτερα ε, τα παράπονα τη κοινότητα Φουλάνη και προσπαθούν να στρατολογήσουν από εκεί. Όμω οι τζιχαντιστικέ ομάδε στην Πουρκίνα και αλλού στην περιοχή περιλαμβάνουν μαχητέ από διάφορε κοινότητε. Ο κίνδυνο για την ασφάλεια δημιουργείται όχι μόνο από την επέκταση των τζιχαντιστών αλλά από τι ε, τι τις ε, υπερβολές και των, ε, των σκοτωμών που λαμβάνουν χώρα με εξοδικαστικό τρόπο. Ο νόμος ε, δίνει τη δυνατότητα σε θέλοντες να βοηθά τις ε, δυνάμεις ασφαλείας και είναι ένας νόμος που υιοθετήθηκε αυτή την εβδομάδα, μπορεί έτσι να κανονικοποιηθούν, αν θέλετε, αυτές οι καταχρήσεις και να βαθύνει η διαίρεση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, αν γίνουν λάθος ε, χειρισμοί. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θυμάται πόσο ε, σημαντική είναι η πολιτική και η διακυβέρνηση, παρόλο που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση ασφαλείας που επιδεινώνεται. Είναι ενθαρρυντικό ότι έχουμε συστάσεις από τη Σύνοδο στο ΠΟ, ότι θα πρέπει η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην απλά εκπαιδεύουν, αλλά να κάνουν και άλλα ε, πράγματα. Γιατί όντως η κατάσταση επιδεινώνεται. Ε, επίσης πρέπει να σας πω ότι η αποστολή PSDC πρέπει να στηριχθεί, αλλά και ευρύτερα να πλαισιώνονται επιτόπου. Είναι κάτι που έχουμε ε, προτείνει εδώ και καιρό. Πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και να ε, ε, βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές να προλάβουν φρικαλαιότητες εναντίον του τοπικού πληθυσμού. Στην Πουρκίνα Φάσο, στο Μαλί, στο, στο Νίγηρα, πρέπει να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν καλύτερα οι δυνάμεις ασφαλείας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Ε, πρέπει να μεταρρυθμιστούν βαθύτερα οι υπηρεσίες ασφαλείας και να ε, μεταρρυθμιστεί και η προσέγγιση που θετεί το κράτος ως προς την ε, διακυβέρνηση. Πρέπει να το γνωρίζει αυτό η διεθνή κοινότητα γιατί η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, είναι εκλογική χρονιά είναι ανάγκη το κράτος να αποδίδει καλύτερα, όχι μόνο να παρέχει υπηρεσίες, αλλά και να κυβερνά πιο ενεργά, καλύτερα και με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί ε, τελικά αυτές οι ομάδες ε, διωγγώθηκαν λόγω της εσφαλμένης διακυβέρνησης των ε, παροηγούμενων καθεστώτων. Σας ευχαριστώ πολύ. είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε για την για την παρουσίασή σας. Όντως είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση. Θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση ασφαλείας, για την περιφερειακή προσέγγιση στο Σαχέλ, για την ανάγκη να έχουμε διασυνοριακή συνεργασία. Η ευρωπαϊκή παρουσία στην Πουρκίνα Φάσο είναι περιορισμένη. Να σας δώσω το λόγο στην κυρία Μάρκουσεν και στη συνέχεια στον αντιστράτεγο Πουλκίνεν. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάτε την κατάσταση, η αποτίμηση της κατάστασης. Τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει, ποιοι είναι οι προβληματισμοί που πρέπει να μας απασχολούν και ποια είναι και τα βασικά εμπόδια. Γιατί υπάρχει δυσκολία να γίνει αποδεκτή μια πιο έντονη ευρωπαϊκή παρουσία. Η κυρία Μάρκοσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε την ανάλυση. Ένα σχόλιο μόνο, αν είναι εδώ ακόμα ο μιλητής μας. Το εθνοτικό ζήτημα είναι σημαντικό και στην Πουλκίνα, Φάσο. Η ανάλυση μας είναι ότι οι Φουλάνοι χρησιμοποιούνται για διαφυλετικές συγκρούσεις. Αλλά αυτό που επίσης διαπιστώνουμε είναι η παράμετρος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Υπάρχουν λίγοι πόροι για τους οποίους αγωνίζονται οι αγρότες. Να πω το εξή ότι από πλευράς Ένωσης υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη προς τον Μπουρκίνα Φάσο. Συχνά όταν μιλάγαμε για Σαχέλ εννοούσαμε Μάλι. Για μας ωστόσο τώρα η Μπουρκίνα Φάσο είναι κομμάτι της προσοχής που δίνουμε. Εμείς ανησυχούσαμε ότι ο πρόεδρος, ένας σοφός άνθρωπος με μακρά πολιτική σταδιοδρομία, αγνοούσε σε κάποιο βαθμό τι μορφή απειλή που αντιμετώπιζε η χώρα. Αυτά ε, άλλαξαν με την αλλαγή του καθεστώτος. Ως Ένωση τώρα κάναμε πολλά και στην αναπτυξιακή συνεργασία και πολιτικά. Έχουμε επενδύσεις από το 2014 μέχρι το 2020 ε, ένα δις ευρώ. Σημαντικό ποσό έχουμε αυξήσει την διαδικασία περιφερειοποίησης εκεί, δηλαδή γίνεται και μια περιφερειακή υποστήριξη της Βουρκίνα Φάσο. Ε, υπάρχει, αν ζητάμε αποτελέσματα, ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι είχαν μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης στην περιοχή, δημιούργησαν κάτι καινούργιο δηλαδή που θα μπορούμε να που, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αλλού. Αυτό το Plan d'urgence pour le Sahel, το πρόγραμμα επίγουσης βοήθειας στο Σαχέλ που θέλουν να μιμηθούμε και για αλλού. Κάτι που δημιούργησαν οι ίδιοι υπουργοί, δικαιο... Ε, υπουργοί οικονομίας της περιοχής για να ενισχύσουν τις δυνατότητες επενδύσεων στις πιο τροτές, στις πιο ευάλωτες περιοχές, που είναι οι βασικές αλλαγές που θέλουν να δούμε διασυνοριακά. Αυτό είναι ένα από τα θετικά. Επίσης, μπορέσαμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των εθνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα στα σύνορα με τον Μπενέ και πόρους και προβλήματα. Επίσης, ενισχύσαμε κάποιες μικτές ερευνητικές ομάδες σε συνεργασία με ε, αεροπορικές δυνάμεις που προγραμματίζουμε για το 2020. Όπως είπα λοιπόν πριν, θέλουμε να εμπλακούμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη. Αυτό που θέλω να πω εν τέλει είναι ότι με την Μπουρκίνα Φάσο θέλουμε να κρατήσουμε την προσοχή, τη δέσμευση της κυβέρνηση, των κυβερνήσεων στις ευάλωτες αυτές τις περιοχές Κάτι που θέλω να πω είναι το εξή. Όταν δουλεύουμε σε θέματα ασφάλειας, πολύ σημαντικό είναι, και το είπαν πολλά κρατημέλη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αν δεν ξέρουμε αν λειτουργεί κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί αν ο, ο τομέας ασφάλειας δεν αντιμετωπίζεται από τον τόπιο πληθυσμό ως πηγή προστασίας, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Η Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής συνδέεται στενά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, άρα θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερη κατάρτιση στον τομέα αυτό. Τελευταίο θέμα. Ο πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, επιτρέπει εκπαίδευση και εξοπλισμό πολιτών για την ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο. Το ξέρουμε, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, αυτοί που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια μας μιλούν για τα προβλήματα της ανθρωπιστικής κατάστασης. Έχουμε 600.000 άτομα που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στον Μπουρκίνα Φάσο. Μεγάλο ποσοστό για μια τέτοια χώρα. Όπως σας είπα υπάρχει επίγνωση των προβλημάτων από την κυβέρνηση και υπάρχουν και τα εργαλεία. Χρειάζεται λοιπόν δράση και από πλευρά τη ηγεσία και από πλευρά του Προέδρου. Ευχαριστώ. Ο στρατηγό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή ήδη ακούσαμε μια διεξοδική παρουσίαση της κατάστασης, από τον πρώτο μας προστεκλημένο. Εγώ θα μείνω σύντομος. Για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις στρατιωτικές της ε, επιχειρήσεις ή δράσεις. Πρώτα απ' όλα για την ε, υποβάθμιση της κατάστασης ασφαλείας. Εγώ από το 2016 που γνωρίζω την κατάσταση βλέπω ότι τα πράγματα αυξάνονται δραματικά. Φαίνεται και από τον χάρτη. Το 2019 μόνο στην Πουρκίνα Φάσο και όχι στο Μαλί είχαμε τεράστια αύξηση. Το βλέπετε και στο χάρτη. Δεν έχουμε μόνο στο βορρά της χώρας πολλούς εκτοπισμένους, αλλά παντού, σε όλη τη χώρα. Χθε, χθε το βράδυ κιόλα, με την επίθεση στο κέντρο της χώρας είχαμε πάλι νεκρούς. Αλλά για την ενημέρωση των στρατιωτικών Ξεκινάμε από τον κόλπο τη Γουινέα, πάμε σε όλη τη ζώνη νοτίω τη Σαχάρα και φτάνουμε στα κέρια τη Αφρική. Μιλάμε για ένα τεράστιο θέατρο επιχειρήσεων. Βεβαίω είναι ένα δρόμο εμπορικό που έρχεται από τον Ατλαντικό και φτάνει ω τη Μεσόγειο στην ουσία, μέσω τη Ερυθρά. Είναι ένα ενιαίο θέατρο αλλά πρέπει να δούμε τα, τα κράτη μεμονωμένα και την περιοχή ως σύνολο το ίδιο. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Έχουμε το πρόβλημα των ε, προσφύγων, των ιστορικών εκτοπισμένων. 500.000 είναι ιστορικώς εκτοπισμένοι. Έχει σχέση αυτό και με τη μεταναστευτική κρίση και είναι δύο οι ομάδες. Η μία είναι η συσχετισμένη με την Αλκάιντα, η και η άλλη με το ΝταΕΣ στην περιοχή της Σαχάρας. Έχουμε πολύ δυνατούς αντιπάλους. Γνωστούς από τη Μέση Ανατολή. Κοιτάζουν να υποδαβλήσουν τα πράγματα λοιπόν και στην περιοχή του Σαχέλ. Και είναι πολύ προηγμένοι στα μέσα που χρησιμοποιούν. Χρειαζόμαστε τις τοπικές δυνάμεις λοιπόν για να προστατευτούμε. Μετά υπάρχει σαφώς σχετισμός μεταξύ τρομοκρατών και εγκληματικών ενεργειών. Δεν λέω βέβαια ότι η εξόριξη χρυσού δεν γίνεται και προς όφελος της κυβέρνησης, αλλά διαμάντια, ελεφαντόδοντο, εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικών, όλα αυτά υπάρχουν εκεί και είναι πηγή χρηματοδότησης για τις τρομοκρατικές ομάδες. Όπως και, όπως και η Μπριζίτ εξήγησε, η κατάσταση μοιάζει με το Μάλι από την άλλη πλευρά των συνόρων στην Πουρκίνα Φάσο. Ιδίως στο κέντρο του Μάλι. Τα σύνορα δεν γίνονται σεβαστά και φυσικά οι τρομοκρατικές δραστηριότητες δεν γνωρίζουν σύνορα. Πάντως, η δική μας επισκόπηση για το πώς είναι η κατάσταση τώρα και πώς μπορεί να εξελιχθεί φέτος, εάν δεν αναλάβουν δράση οι ίδιοι κάτοικοι της Μπουρκίνας και δεν υποστηριχθούν από τη διεθνή κοινότητα, θα καταρρεύσει όλη η κατάσταση. Τώρα για τις εντολές των επιχειρήσεων της Ένωσης και την παράταση στην Μπουρκίνα Φάσο, έχουμε ήδη ξεκινήσει να το συζητάμε. Μέχρι τώρα μπορεί η επιχείρηση του Μάλι να, να προσφέρει και στην Μπουρκίνα μια προστασία ως παρακλάδι χάρη στην ομάδα του Σαχέλ, τον G5. Δεν έχουμε όμως δικό μας νομικό σύμβουλο στα επιτελεία αυτά. θα πρέπει να στείλουμε ομάδα για εκπαίδευση και στην Πουρκίνα Φάσο όπως και στο Μάλι. Και ήδη από το Μάλι έχουμε, λάβει, έχουμε μάθει κάποια πράγματα Θέλαμε να, ε, Ήθελα να σχολιάσω στη σύντομη παρουσίασή μου το θέμα του... της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, αλλά πώς είναι διοργανωμένες οι δυνάμεις στο Μάλι και στην Μπουρκίνα Φάσο. Είναι πολύ εκτεθειμένοι. σε περιπτώσεις χτυπημάτων που είναι θανατηφόρα. Μπορεί να χάσουν και το 100 ή το 99% των ε, δυναμεών τους. και γιατί δεν είναι σωστά διαρθρωμένοι. Οι μονάδες πρέπει να έχουν καλύτερη σύνθεση, να είναι μεγαλύτερα τα σταταύματα, να μπορούν να αυτοπροστατευτούν σε πρώτη φάση και να κοιτάξουν και τα σύνορά τους. για το τι μπορεί να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αποστολή της εκπαίδευσης. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να διευρύνουμε την εντολή για να καλυφθεί εκτός από το Μάλι Φάσο και να δούμε τι παρουσία μπορεί να έχουμε στη Γουαγκαντούγκου ή και αλλού. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η άλλη είναι να χειριστούμε την Μπουρκίνα με έδρα τον Παμάκο, την Παμάκο, με την έγκριση βεβαίως της κυβέρνησης της Μπουρκίνας. Συμβουλευτικά τουλάχιστον πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους. Πρώτα απ' όλα ο Αγνόντον Ζων για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε ζωφερή εικόνα, δεν μας εκπλήσει. Και κάπως ευνηδιαστήκαμε βέβαια εκεί που δεν περιμέναμε να πάρουν αυτή την τροπή τα πράγματα. Ξέραμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι μπορεί να υπάρξει επαναχώρηση, αλλά μπήκαμε πάλι σε ε, μια ελικοειδή πορεία ε, που είναι ατυχής παρά τις οικονομικές προσπάθειες που έχουν γίνει και οι ευθύνε είναι πολλών. Δεν θέλω βεβαίω να απαλλάξω από καθευθύνη τις τοπικές αρχές, γνωστή η κατάσταση, αλλά έχω μία ερώτηση για τον Άντου. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ταμπού στην όλη περιοχή. Μιλάμε για ομάδα τσιχαντιστών. Πολλές κυβερνήσεις, πολλές από τις τοπικές αρχές. Επί χρόνια συζητούσαν με ομάδες τζιχαντιστών για να μείνουν εκτός των χωρών τους. Μπουργκίνα, το ξέρει ο κόσμος όλος, είχε αυτή την πολιτική ε, υπό τον προηγούμενο πρόεδρο. Με ένα μπλεγμένο δίκτυο, όμως είχε πετύχει τη σταθερότητα βρίσκοντας τρόπους συνεννόησης με διαφορετικές ομάδες. Εγώ ήθελα να καταλάβω σε τι βαθμό σήμερα η υποβάθμιση τη κατάσταση, η εκτραχύλιση της κατάσταση στην Μπουρκίνα έχει σχέση με τα εσωτερικά τη χώρας, πρώτον και δεύτερον, χωρίς να παραβλέπουμε την αποφασιστικότητα και επιθετικότητα των ομάδων των τζιχαντιστών, διότι ακόμη και αν μπορούν να διαβρώσουν κάποιες κοινότητες και να τις δείσουν εκεί με το λαθρεμπόριο, με την εμπορία, ιδεολογικά έχουν ένα πρόγραμμα προσελητισμού, έχουν στρατηγικό σχεδιασμό να, εγκαταστα... να εδρεωθούν σε κάποιε περιοχέ και να τι αποσταθεροποιήσουν. Μην το παραβλέπουμε αυτή την παράμετρο, αλλά ε, σίγουρα κάποιε ε, αναταραχές που υπήρχαν εσωτερικώ στην Πουρκίνα μπορούσαν να τι εκμεταλλευτούν. Μήπω είναι αυτό ένα λόγο. Ευχαριστούμε η κυρία Κάγκο για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ κύριε Λουαζό. Είναι πολύ συγκριτικό να ακούω να συζητιέται η κατάσταση στην Πορκίνα Φάσο και στο Σαχέλ εν γέννη. Όχι μόνο γιατί από εκεί έρχομαι, αλλά γιατί καταλαβαίνω τις διαστάσεις του προβλήματος. Ευχαριστώ τον κύριο Ντανζό για την έκθεση που συνέταξε. Έχουμε υποβάλει μια μικρή τοπολογία για την Πορκίνα Φάσο που έγινε δεκτή και σας ευχαριστούμε. Και θα συνεχίσω στα αγγλικά για να τιμήσω και την ε, πολιτική μου ομάδα που δεν είναι γαλλόφωνη. Έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Πρώτον, στην κυρία Ράσμουσεν. Λέτε ότι έχουμε 600.000 εσωτερικώς εκτοπισμένους. Αυτό για μια τόσο μικρή χώρα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά ίσως θα μας, μπορούσατε να μας δώσετε ιδέες για το πώ να το χειριστούμε καλύτερα. Και μετά μιλήσατε για το πόσο σοβαρέ είναι οι επιπτώσει τη φτώχεια. Μπορείτε να μα πείτε και εδώ κάτι παραπάνω. Ποια είναι η εξέλιξη από το αντίκτυπο τη φτώχεια, γιατί πάντοτε ήταν μια πολύ φτωχή χώρα η Μπουρκίνα, ακόμα και πριν αρχίσουμε να μιλάμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έχετε δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχει συσχετισμό και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς έχει μετεβληθεί η κατάσταση εκεί. Και μετά μια δεύτερη ερώτηση για το στατικό. Με συγχωρείτε, μου διαθέτει το όνομα. Ε, είπατε ότι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την κατάσταση στο Μάλι. Πρώτο σχόλιο να πω ότι από την δική μου εμπειρία και από όσα έχω ήδη ακούσει, οι Γάλλοι βρέθηκαν ε, τελείως μόνοι στο Μάλι. Και ακόμη και όταν το συζητάμε εδώ στο Ευρωβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση στο Σαχέλ, στην Μπουρκίνα Φάσου. Εγώ είχα επισκέπτε μια ομάδα φοιτητών την περασμένη εβδομάδα και ένα με ρώτησε. Δεν είναι πατερναλιστικό να πηγαίνουμε εκεί και να του λέμε τι να κάνουν. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε την, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα, ότι πάμε εκεί να ξαναχτίσουμε τα κράτη και να επικεντρωθούμε στη διάσταση της ασφάλειας. Δεν ε, είναι το ερώτημα αν πρέπει κάτι να κάνουμε ή όχι. Βεβαίω και πρέπει, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο πόσα συμβαίνουν. Αλλά για την Πουρκίνα Φάσο είναι χώρα ε, που βρίσκεται πολύ κοντά στις χώρες του Σαχέλ. Έχουμε τώρα ομάδες τζιχαντιστών να δρούν εκεί και πρέπει εμείς η Ευρώπη να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, να καταγγείλουμε από τι ομάδε των τσιχαντιστών. Ο Καμί νομίζω είχε πει ότι όταν δεν πει τα πράγματα με το όνομά του, δεν μπορεί ποτέ να βρει και λύση. Α έχουμε λοιπόν αυτό το θάρρο και η συγκεκριμένη μου ερώτηση προ εσά είναι όταν λέτε ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα από το Μάλι και πώς να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, λέτε τα εισοδήματα από την εξόρυξη χρυσού χρησιμοποιούνται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από κλιματικές ομάδε. Τι εννοείται ακριβώ, μπορείτε να το εξηγήσετε. Και το γεγονό ότι κάποιε εταιρείε ε, ε, που έχουν ασχοληθεί με την εξόρυξη του χρυσού θα μπορούσαν να δώσουν θέσει εργασία και εισόδημα. Αυτό ήταν σημαντικό για τον προπολογισμό μια χώρα όπω η Μπουρκίνα. Και για να κλείσω, πώ θα το εξορροπήσετε αυτό, πώ θα το αντισταθμίσετε ε, και πώ θα υλοποιήσετε ακριβώ αυτό που ανέφερε και η πρόεδρο. δεν είναι τόσο εύκολο να προστατευτούν τα ορυχεία αυτά. Και ο κόσμος που ζει εκεί μπορεί να βρεθεί να απειλείται. Και μετά το θέμα των γυναικών, ε, εξίσου σημαντικό. Ξέρουμε τι κάνουν οι τζιχαντιστέ οι γυναίκες εκεί που έχει διεγκωθεί το φαινόμενο. Έχουμε τη σχετική εμπειρία στη Συρία, το Ιράκ. Ξέρουμε πώς, ε, επισφαλή είναι συνηθίσει των γυναικών. Μα ανησυχεί πολύ λοιπόν τι έχετε παρατηρήσει στην πράξη, τι συμβαίνει ω προ τη διάσταση αυτή, την έμφυλη. Ευχαριστούμε για του Renew Europe, ο κύριος Αστρεβίτσιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από όλες τις πληροφορίες που μας δίδεται, είναι σαφές ότι η τάση αποσταθεροποίησης ε, είναι αυξητική. Το 2019 ήταν ε, το έτος ε, όπου κορυφώθηκαν ε, οι θάνατοι, οι επιθέσεις, οι ανθρώπινες απώλειες, το γεγονός ότι ολόκληρες περιφέρειες και περιοχές κατέλαβαν οι ένοπλες ομάδες και το καθεξής. Δεν βλέπω άλλη τάση. Ο κύριος Πουλκίνεν ήταν σαφές, σαφής στην τοποθέτησή του. Άρα, εάν δεν ε, δράσουμε έγκαιρα, θα αποτελέσουμε μέρος της δυστυχούς διαδικασίας και του χρόνου θα συναντηθούμε εδώ για να απαριθμίσουμε ακόμα μεγαλύτερα νούμερα, ακόμα πιο αρνητικές ε, επιπτώσεις και ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις που θα έχουν καταληφθεί από τους αντιπάλους μας. Εάν ε, ε, δεν ε, προχωρήσει η αποστολή CSTP, ποια θα είναι η εναλλακτική, τι θα κάνουμε, απλά θα κάνουμε καταγραφή των στατιστικών, μήπως πρέπει να δράσουμε έγκαιρα. και να λάβουμε αποφάσεις οι οποίες επίγουν. να μην στηρίξουμε απλά το λαό και τη χώρα με τις πολιτικές δηλώσεις και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση και αν δεν αναλυφθεί δράση, ποιες είναι οι Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, από την περιγραφή που κάνετε από την κατάσταση και από εσάς αλλά και από τον προσκεκλημένο μας μέσω Skype, ε, μου δημιουργείται στο μυαλό το εξής ε, ερώτημα. Διαφαίνεται ότι θα καταρρεύσει το κράτος, το κεντρικό, οι βασικές αρχές. Πόσο μέρος της χώρας ε, ε, ελέγχει τελικά η κεντρική κυβέρνηση, το επίσημο κράτος. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι να καταρρεύσει πλήρως. Πληρώνονται π.χ. οι μισθοί στις αυτόνομες περιοχές. Υπάρχει γενική αποσύνθεση των βασικών δομών του καράτους. Είναι κάτι πολύ υπερβολικό να ισχυριστεί κανείς ότι διαλύεται το κράτος στη χώρα αυτή και οι κρατικές δομές. Αν υπήρχε πολιτική βούληση και αν υπήρχαν και οι απαραίτητοι ε, πόροι, Μήπως θα πρέπει να στηρίξουμε και να είμαστε παρόντες ως ευρωπαϊκές χώρες και ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να αποθήσουμε όλους αυτούς τους τσιχαντιστές. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τελικά πόσα χρειάζονται, τι χρειάζεται. Και αν δεν είμαστε σαφείς για το πώς μπορεί να πετύχουμε κάτι τέτοιο, και πώς μπορούν να ε, εξουδετερωθούν αυτές οι δομές. Αν δεν μιλήσουμε ξεκάθαρα για το τι χρειάζεται για να τις εξουδετερώσουμε αυτές τις δομές, ε, δεν θα έρθουν αποτελέσματα, όπως το είπαν και οι προλαλήσαντες, όπως το είπε και η Πέτρα. Μπορεί να περιγράφουμε την κατάσταση, όπως το είπε και ο Πίτερ, ο κ. Στρεβίσιος. Ίσως δεν είναι πολύ δημοφιλές να στείλει κανείς στρατεύματα στην Μπουρκίνα Φάσο, αλλά μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί και να, αφήσουμε, να επιτρέψουμε στους άλλους να αναλάβουν τον έλεγχο όλης της περιοχής και της χώρας. Μπορεί να είναι αυτή μια απάντηση. Άρα να αξιολογήσουμε πόσες δυνάμεις έχουν μείνει στο κράτος της Μπουρκίνα Φάσο πάνω στις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε και τις οποίες μπορούμε να ενισχύσουμε. Καταρχάς. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ο Σβέν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθώ, παρεμφερεί είναι τα ερωτήματά μου. Όντως η αξιολόγηση της κατάστασης ε, ε, γίνεται με πολύ δυσάρεστο τόνο και δυσάρεστη χρειά. Έχουμε τζιχαντιστές, τρομοκρατικές ομάδες και το καθεξής. Μετά βλέπουμε την αποστολή CSDP και έχουμε εκπαιδευτική αποστολή η οποία μάλιστα λειτουργεί με έδρα το Ουαγκαντούγκου. Λίγο είναι αυτό το εκπαιδευτικό στρατιωτικό σκέλος, δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος της πρόκλησης. Είστε αισιόδοξοι, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει απόφαση να αναπτύξει μια τέτοια αποστολή κανονικά στρατιωτική στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να αντιστρέψει αυτό τον ρου των πραγμάτων, μπορεί να αντιστρέψει την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην ευρύτερη χώρα και αν είναι δύσκολο να αντιστραφεί η πορεία των πραγμάτων, θα μπορέσει αυτή η αποστολή ακόμα και αν την αποφασίσουμε να φέρει σταθερότητα στη χώρα. Και μιλούμε για απαιτούμενη βοήθεια, αλλά σε ποιο μέγεθος, πόση ακριβώς για να μπορέσουμε να ε, ε, αναχαιτήσουμε αυτή την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας. Χρειάζονται επιχειρήσεις σε ποια κλίμακα για να ε, πετύχουμε κάτι ή για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Να, κάνουμε, να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές μας, στον καθένα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Πρώτα στον αντιστράτηγο Πούλκινον, στη συνέχεια στην κυρία Μαρκούσεν και τελευταίος ο κύριος Λέμποβιτς που μίλησε πρώτος στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι εξαιρετικά τα ερωτήματά σας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ολοκληρωμένες απαντήσεις, εμπεριστατωμένες. Γιατί κάποιες από τις δηλώσεις μου είναι, ε, έχουν χαρακτήρα πρόβλεψης. ξεκινώντας από το σύνδεσμο τη σχέση μεταξύ εγκληματικότητας και ισλαμιστικών ομάδων. Είναι μία πρόβλεψη, μία εκτίμηση, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχουν και υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ εγκληματικότητα και ισλαμιστικών ομάδων, όχι μόνο στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικά. Μπορεί αυτό είναι ένας λόγος για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας και όντω οι τζιχαντιστές έχουν ενδιαφέρον να ασκούν, να διαπράττουν εγκληματικές δραστηριότητες γιατί αυτό αυξάνει ε, τις ε, προσόδους τους, τα έσοδά τους. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, παρόλο που είναι εκτίμηση αυτή, έτσι, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας στην Μπουρκίνα Φάσο. Αν δείτε τη δική μου εντολή, την εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι είναι μη εκτελεστική. Δηλαδή, πρέπει να παραμείνουμε στα της εκπαίδευσης. Πρέπει να παραμείνουμε σε ένα ρόλο καθαρά συμβουλευτικό και έμεσο και να μην εμπλεκόμαστε σε καμία επιχείρηση άμεσα, σαν παράγοντες, σαν πρωταγωνιστές. Οι τοπικές αρχές πρέπει να το κάνουν αυτό και αυτή είναι η διαφορά της άμεσης από την έμεση ε, παρέμβαση και παρουσία. Αυτό καταρχάς. Κάτι άλλο που ανέφερα είναι το εξής. Την έμφαση στην εκπαιδευτική αποστολή. Χρειάζεται να πλησιάσουμε, να είμαστε πιο κοντά στις δομές και να αναπτύξουν κρατικές αρχές ε, δομές με τρόπο αξιόπιστο. Εκτίθενται τώρα στις ε, τζιχαντιστικές ομάδες οι οποίες έχουν πολύ προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες. Είναι μια διαδικασία αυτή που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φέρνει καρπούς σε βάθος χρόνου, αλλά δεν ανταποκρίνεται και δεν ταιριάζει ε, σε περιόδους όπου η κρίση είναι οξυμένη, ε, σε περιόδους όξυνσης, ε, σε βραχυπρόθεσμα. Επειδή πρέπει να συμφωνούμε 26-27 χώρες, δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι όσο μια μικρή συμμαχία. Παρ' όλα αυτά πολλά μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δρά ε, ομοφόνος σιγά σιγά. Ε, τώρα, για να, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι, να προλάβουμε την κατάραψη της κυβέρνησης, τότε θα προλάβουμε η κυβέρνηση, ε, το κράτος ε, της Μπουρκίνα Φάσο ε, να διατηρηθεί. Το ίδιο έκανε και η Γαλλία πριν από 10 χρόνια και κατάφερε να διατηρηθεί το κράτος του Μαλή. Έχουμε νομικά μέσα, έχουμε οικονομική παρέμβαση, οικονομικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το βασικό όμως είναι η αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό και από, κυρίως από την κυβέρνηση διστάζει η κυβέρνηση να δεχθεί τη στήριξή μας. Ίσως έχει αρνητικό προηγούμενο, δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ε, ξεπεράσουμε. Ίσως τα ήπια στοιχεία άσκησης εξωτερικής πολιτικής θα φέρουν περισσότερα αποτελέσματα από ε, μια ακαθαρά στρατιωτική χειρή παρουσία. Μπορεί και όχι, δεν το αποκλείω. Είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Συμφωνώ με όλους εσάς. Πρέπει περισσότερα πράγματα να κάνουμε και για την παροχή συνθήκων ασφαλείας. Πρέπει να επανεξετάσουμε την εντολή μας και τη στήριξη που δίνουμε στην Πουρκίνα Φάσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κύριε Μάρκουσεν. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Αν υπάρχει διάλογος με τις ένοπλες δυνάμεις και τον τοπικό πληθυσμό στην περιοχή. Ο πρόεδρος Καμπορέ είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα είχε την ίδια συνεργασία που είχε ο Μπλέζ ωραίο ο προηγούμενος πρόεδρος αλλά υποστηρίζει τις διαδικασίες που είναι υπό εξέλιξη σε κάποιες περιοχές. Αλλά η επίσημη θέση είναι αυτή. Αυτή είναι η άποψη του Καπορέ για τους 600.000 εσωτερικά εκτοπλισμένους και τις αιτίες Καταλαβαίνω ότι έχετε σχέσεις με την περιοχή, συγγενείς εκεί. Οι 600.000 άνθρωποι ε, παίζουν ένα ρόλο. 18 ε, εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι της χώρας. Μισό εκατομμύριο είναι μεγάλο ποσοστό. Η ΕΚΟ έχει παρέμβει και αύξησε την παρέμβασή της εκεί, αλλά οι εσωτερικά εκτοπισμένοι μπορεί να μένουν ε, με οικογένειες, αλλά είναι οικογένειες επίσης φτωχές, δηλαδή δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ξεκινήσει μία μελέτη της φτώχειας εκεί. Δεν έχουμε τα στοιχεία ανάπτυξης τα τελευταία, αλλά ο αριθμός των επιθέσεων και ο βαθμός ανασφάλειας σίγουρα θα επηρεάσουν την περιοχή. Αν υπάρχει κατάρρευση, ήταν η τελευταία ερώτηση, υπάρχει κατάρρευση της κυβέρνησης του κράτους, τι πιθανότητες ε, υπάρχουν. Καταρχάς, εμείς κάναμε σημαντικά κομμάτια ανάλυσης για το ρόλο της Ένωσης σε πολλές, για πολλές από αυτές τις χώρες αν δεν υπήρχε μια ισχυρή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Εμείς παίξαμε σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν σε λειτουργία συστήματα. Αυτό που πρόκειψε από, την, ε, από τις έρευνές μας είναι ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Είναι σοβαρό το θέμα λοιπόν. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε με πολλές πρωτοβουλίες είναι εν ώψη της διάσκεψης 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες είναι να δουλέψουμε για την ανάλυση αναγκών και ανάλυση κενών ούτως ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα τι λείπει, τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς και οι χώρες σε τομείς σταθεροποίησης και για περιφερειακή διάσταση και για τομείς. Αυτό, που, αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ως Ένωση. Ο ύπατος εκπρόσωπος είπε ότι ήρθε η στιγμή να κλιμακώσουμε την παρέμβασή μας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να κλιμακώσει την παρέμβασή της. Ευχαριστώ. Κύριε Λέμποβιτς. Κάνα δύο ερωτήσεις. Ένα, η πολιτική ανακατάταξη και ο αντίκτυπό τη. Η Μπουρκίνα Φάσο δεν είναι η μόνη χώρα όπου υπάρχουν καταγγελίες για συνεργασία της κυβέρνησης με τζιχαντικιστές και για το Μάλι υπάρχει αυτή η αντίληψη και τον πρόεδρο του ΡΕ. Πάντως η εμπλοκή του, της στρατιωτικής ηγεσία και των τζιχαντιστών είχε έναν αντίκτυπο στην δυσχέρανση του να μπορέσει να απαντήσει η χώρα στην αύξηση της τζιχαντικής παρουσίας. Αλλά οι διαπραγματευτές, αυτοί με τους οποίους διαπραγματευόταν ε, η Βουκίνα Φάσο το ρώ και το 13, δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε με την υποστήριξη κάποιων από την κυβέρνηση, όχι όμως πάντα των ίδιων και όχι πάντα των ε, φορέων εκείνων οι οποίοι είχαν εμπλακεί στο ξεκίνημα της δραστηριότητα. The counter coup uh, that happened in Burkina Faso did play a role, but again, I, I really want to emphasize that these um, these arrangements that were in place